Good afternoon, Καλώς ορίσατε. Θα αρχίσουμε τη συνεδρίαση στην Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών. Έχετε όλοι λάβει το σχέδιο μέσα διάταξης. Υπάρχουν σχόλια παρακαλώ. Όχι, από ό,τι βλέπω. Άρα εγκρίνεται. Και περνούμε στο σημείο 2. Ανακοινώσεις του Προέδρου. Μπορείτε να μιλήσετε βουλγαρικά, τσεχικά, δανικά, γερμανικά, ελληνικά, αγγλικά, ισπανικά, φινλανδικά, γαλλικά, ουγγρικά, ε, λιθουανικά, τέλος πάντων διάφορες γλώσσες μεταξύ των οποίων και τα ελληνικά. Ελπίζω να σας φτάνουν αυτές οι γλώσσες. Αν σα έρθει να μιλήσετε σε κάποια άλλη γλώσσα, καλή τύχη, δεν σα σας καταλάβει κανένας. Αλλά θα πρέπει να ξέρετε πώς αναμεταδίδεται ζωντανά η συνεδρίαση στο διαδίκτυο αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Καλωσορίζω τον κύριο Μόρο Ολιβιέρα Είναι εδώ. από τη γραμματεία. Περνούμε τώρα στο σημείο 3, το βασικό δηλαδή θέμα της συνεδρίασής μας, ακρόαση με θέμα η απαλλαγή που χορηγείται στους αποκεντρωμένους οργανισμούς, διακυβέρνηση και λειτουργική αποτελεσματικότητα. Έχουμε διάφορους προσκεκλημένους, μεταξύ των οποίων και κάποιοι βουλευτές. Θα ήθελα να ακούσουμε πρώτα τον ε, εισηγητή που θα μας κάνει την εισαγωγή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, Αντιπρόεδρε, τη σε επιτροπή, σε αγαπητοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας καλωσορίσω στη σημερινή μας ακρόαση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα. Πρόκειται για χορήγηση απαλλαγή στους αποκεντρωμένους οργανισμούς, διαχείριση και λειτουργική αποτελεσματικότητα. Όλος ιδιαίτερος θα ήθελα να καλωσορίσω τους προσκεκλημένους που μετέχουν στη σημερινή δημόσια ακρόαση. Την έχουμε καταμερίσει σε τέσσερα τμήματα όπως βλέπετε και στο ημερήσια διάταξη τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιήθηκα ενεργά στον τομέα των αποκεντρωμένων οργανισμών. Ήμουν εκπρόσωπος των σοσιαλιστών για τη διαδικασία απαλλαγής του 2008 και κατόπιν η για 22 αποκεντρωμένους οργανισμούς και 5 κοινοπραξίες για το ε, οικονομικό έτος 2009. Ε, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η εμπειρία και έχω αποκομίσει μεγάλη εμπειρία. Τα τελευταία χρόνια λοιπόν συναντήθηκα με τους διευθυντές όλων των αποκεντρωμένων οργανισμών, μετέβην και επιτόπου σε διάφορους οργανισμούς για να διαπιστώσω πώς λειτουργούν επιτόπου. Πλούσια εμπειρία και αυτή η στενή συνεργασία ενίσχυσε την πεποίθησή μου ότι οι αποκεντρωμένοι οργανισμοί αποτελούν προσθέμενη αξία για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ενισχύουν περαιτέρω την ευρωπαϊκή ταυτότητα με την επιτόπου παρουσία στα κράτη-μέλη επί σειρά ετών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εποπτείας στα πλαίσια πάντοτε της χορήγησης απαλλαγής το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε την ευκαιρία να ξεκινήσει ένα επικοδομητική διάλογο με τους αποκεντρωμένους οργανισμούς με το εσωτερικό, την εσωτερική υπηρεσία ελέγχου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και με το ελεγκτικό συνέδριο. Όλη αυτή η ενδελεχής εργασία κατά τη γνώμη μου οδήγησε σε αυξημένη διαφάνεια καθώς και σε αυστηρότερη ε, διαχειριστική πειθαρχία. Ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό είναι αυτό της ΣΥΠΟΛ ε, πέραν κάθε αμφιβολία ε, υπό τη διοίκηση του νέου διευθυντή, η ε, ΣΑΙΠΟΛ κατάφερε να διορθώσει διάφορες παρατυπίες που έπληκταν τον οργανισμό τα τελευταία χρόνια παρόλα. Αυτά κανεί δεν μπορεί να αρνηθεί το ότι αυτή η βελτίωση τη αποτελεσματικότητα στη διαχείριση τη ΣΑΙΠΟΛ οφείλεται μεν σε αυτή την κατεύθυνση αλλά και στην πίεση που άσκησε η Επιτροπή μας για να αντιμετωπίσει και να δώσει μια απάντηση ή να ρυθμίσει τις εντοπιστείς σε παρατυπίες. Ευελπιστώ ότι η να ρυθμισει τις εντοπιστησεις παρατυπίε. παρατυπιες ευελπιστω οτι η διαδικασια χορηγησης απαλλαγης ε, για τους οργανισμούς για το 2010 θα χαρακτηριστεί από έντονες προσπάθειες όλων των εμπλεκόμενων φορέων και θα καρποφορήσουν αυτές οι προσπάθειες ούτως ώστε να έχουμε καλύτερα σε σχέση με το παρελθόν αποτελέσματα. Αληθεύει ότι η διακήρυξη ε, ε, και η λειτουργική αποτελεσματικότητα είναι θέμα που που ε, κατήχε προεξάρχουσα θέση ε, σε διάφορες ε, εκθέσει τη Επιτροπής μας για τη χορήγηση απαλλαγή σε διάφορου αποκεντρωμένους οργανισμού. Τα τελευταία χρόνια, στα πλαίσια τη διαδικασία απαλλαγή, αυξάνεται διαρκώ το, ο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το θέμα τη ηλεκτρονική διακυβέρνηση ήταν στον πυρήνα των συζητήσεων και διαφόρων μελετών. Η Επιτροπή Ελέγχου των προπολογισμών, επίση τα πεπερασμένα χρόνια εκπώνησε μία έκθεση πρωτοβουλία με οριζόντιου χαρακτήρα παρατηρήσει σχετικά με ατέλειες, προκλήσει και τι βέλτιστε πρακτικέ σε σχέση με του αποκεντρωμένου οργανισμού, πέραν από την απόφαση χορήγηση απαλλαγή για κάθε μεμονωμένο οργανισμό. Σε κάθε μία από αυτέ τι εκθέσει από του μεμονωμένου οργανισμού, καθώ και σε αυτή την έκθεση πρωτοβουλίας που προανέφερα βλέπουμε ε, πλήστα παραδείγματα βελτίστων πρακτικών καθώ όμω και ατέλειε και δυσλειτουργίε που εντοπίσαμε επίσης προτάσεις ε, για να ε, βελτιώσουμε τη διαδικασία. Μέσα σε αυτή την έκθεση ε, σχολιάστηκαν λοιπόν θετικέ και αρνητικέ πτυχέ τη οικονομική διαχείριση, το θέμα των ανθρωπίνων πόρων, ε, τα εσωτερικά συστήματα ελέγχου και ευρύτερα ζητήματα διακυβέρνηση. Ε, δύο βασικοί εταίροι τη Επιτροπή μα πρότειναν τρόπου βελτίωση τη διαδικασία και αναβάθμιση αποτελεσματικότητα. Πρόκειται για την διαθεσμική ομάδα εργασία για του αποκεντρωμένου οργανισμού καθώ και το ελεγκτικό συνέδριο. Από αυτή την πλευρά πλευρά προσμένω με ανυπομονησία την ε, συνεισφορά τη ε, διαθεσμική αυτή ομάδα εργασία για του αποκεντρωμένου οργανισμού. Τρία από τα διακεκραμένοι μέλη τη εξάλλου θα μα παρουσιάσουν ε, του τρει διαφορετικού αποκεντρωμένου οργανισμού. Είναι εδώ μαζί μα και περιμένουμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον την έκβαση των συζητήσεων στην ομάδα και όλο ιδιαίτερο ω προ τι προκλήσει στι οποίε καλούνται να αντεπεξέλθουν οι αποκεντρωμένοι οργανισμοί. Επιπλέον, το ελεγκτικό συνέδριο έχει αναλάβει και διεξάγει τώρα μία ενδελεχή ανάλυση σε σχέση με την ορεινή κατάσταση όπου ενδέχεται να ανακύψει σύγκρουση συμφέροντων ως προς τους αποκεντρωμένους οργανισμούς. Ε, προσβλέπουμε στην περάτωση αυτή τη ανάλυση και την υποβολή τη σχετική έκθεση στην Επιτροπή μας. Ε, επίσης, ε, περιμένουμε τις εκθέσεις σχετικά με του αποκεντρωμένου οργανισμού που τώρα εξετάζονται από το ελεγκτικό συνέδριο. Θα ήθελα να τονίσω πόσο σημαντικό είναι ο ρόλο του ελεγκτικού συνεδρίου ανέκαθεν δεν ήταν στη διάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και οι εκθέσει του υπήρξαν ένα πολύτιμο εργαλείο στη διαδικασία ελέγχου του Κοινοβουλίου. κλείνοντα. θα ήθελα να τονίσω πω η Επιτροπή Ελέγχου των προπολογισμών θα έπρεπε να ενισχύσει την περαιτέρω τη συνεργασία τη με αυτού του επαγκεντρωμένου οργανισμού. Θέλουμε να προσφέρουμε την υποστήριξη, την καθοδήγησή μα και να καταθέσουμε συστάσει για να συμβάλλουμε και εμεί στην αναβάθμιση τη αποτελεσματικότητα των τον οργανισμό. Θα βάλω μία τελεία εδώ. Θα κλείσω την, παρουσία, την εισαγωγική μου παρουσίαση. Πρόεδρε, σας παρακαλώ, ε, μπορείτε να δώσετε το λόγο στους προσκεκλημένους ε, και στα μέλη της Επιτροπής. Σας ευχαριστώ πολύ. Μετά από αυτή την ε, γενική εισήγηση θα ήθελα να προχωρήσω στο πρώτο τμήμα της σημερινής ακρόασης και θα ήθελα να καλωσορίσω τον κύριο Οσί μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου της Αν Γένσεν. Σας καλωσορίζω, καθώς και τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τέλος, τον εκπρόσωπο του Συμβουλίου, γιατί θα θέλαμε να γνωρίζουμε και την άποψη του Συμβουλίου. Δίνω το λόγο στον κύριο Οσή, μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μπορείτε να μιλήσετε για 20 λεπτά περίπου. Με μεγάλη χαρά βρίσκομαι εδώ σήμερα με τους συναδέλφους σας για να συζητήσουμε αυτό το θέμα που αφορά την συνεργασία των διαφόρων υπηρεσιών. Βρισκόμαστε σε μια χρηματοπιστωτική κρίση η οποία δεν υποχωρεί και ξέρουμε ότι υπάρχει διαθεσμική δέσμευση για να συζητήσουμε θέματα που αφορούν την αξία των χρημάτων μας, δηλαδή το αντίτιμο που οφείλουμε να λάβουμε. Υπάρχουν 40 γραφεία και υπηρεσίες εκτελεστικού χαρακτήρα, ε, έχουν έσοδα 1,7 δις ευρώ, απασχολούν 8.000 πρόσωπα και αυτό έχει μεγάλη σημασία μέσα στα πλαίσια του διοικητικού προϋπολογισμού, του προϋπολογισμού διοικητικών δαπανών. Έχω αναλάβει αυτό το χαρτοφυλάκιο εδώ και ένα χρόνο. Και ρωτώ, θα δαπανούσα δικά μου χρήματα κατά αυτό τον τρόπο. Μπορώ, μπορούμε να βοηθήσουμε ώστε να λειτουργήσουν καλύτερα αυτές οι υπηρεσίες και τα γραφεία, έτσι ώστε να ε, λειτουργούν καλύτερα. Είχα και πρόθεσα πολλές επισκέψεις και με τον κύριο Σεύκοβιτς και όπως είπε και ο κύριος Σταυρακάκης μας ενδιέφερε επιτόπου να δούμε πώς εργάζονται αυτές, αυτοί οι φορείς. Επίσης αυτό έγινε και με τη συνεργασία του Κοινοβουλίου και επίσης στο ελεγκτικό συνέδριο διενεργούνται δύο μελέτες ως προς το benchmarking καταρχήν. Για το benchmarking βρισκόμαστε στο 17ο προσχέδιο. Είχαμε πολύ καλή συνεργασία με τους επιτρόπους με επικεφαλής τις 22 αυτές υπηρεσίες και οργανισμούς. Ήταν μοναδική ευκαιρία για τα μέλη αυτής της Επιτροπής να εκφράσουν τις απόψεις τους. Και έτσι θα μπορέσουμε να λάβουμε υπόψη την ε, άποψη όλων των θεσμικών οργάνων. Θα ήθελα με την άδειά σας να συζητήσω τρία ζητήματα. Καταρχήν την διακυβέρνηση, τη συνεργασία και τους προϋπολογισμούς. Ως προς τη διακυβέρνηση, λαμβάνουμε υπόψη ότι ένα διοικητικό συμβούλιο δεν είναι το μόνο μέσο δράσης γιατί πολλά διοικητικά συμβούλια παρτίζονται από 19 μέλη. Ο μέσος όρος είναι 47 άτομα. Συνέρχονται τρεις φορές το χρόνο μόνο. Οι οργανισμοί είναι αυτόνομοι και έτσι δημιουργήθηκαν. Πιστεύω ότι στον δημόσιο τομέα, εάν υπάρχει αυτονομία, τότε υπάρχει και επάρκεια. Γνωρίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέβαλε προτάσεις για ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης το οποίο να είναι διτό. Να έχουμε το ευρύ διοικητικό συμβούλιο αλλά και μία νέα διαστρωμάτωση εκτελεστικού χαρακτήρα διακυβέρνησης έτσι ώστε να έχουμε ένα μακρόπνο σχέδιο για τους οργανισμούς αυτούς. Ως προς τη λειτουργία τους, εμείς αναρωτηθήκαμε στο ελεγκτικό συνέδριο ως προς το προσωπικό, ποιο μέρος του προσωπικού ασχολείται με καθαρά διοικητικό έργο. Είναι πολύ δύσκολο να το απαντήσουμε, διότι η οριοθέτηση μεταξύ διοίκησης και ε, λειτουργικών εξόδων είναι κάτι ε, το πολύ δύσκολο. Υπάρχει προσωπικό που ασχολείται καθαρά με διοικητικά θέματα, δηλαδή ανθρώπινο δυναμικό, ανθρώπινη πόρη και ούτω καθεξής. Συνολικά, ένα 22% του προσωπικού ασχολείται αποκλειστικά με, διοικητικά, ε, με διοικητικό έργο και πολλές φορές υπάρχει ένα φάσμα μεταξύ 12 και 36% απασχόλησης. Αλλά αυτό δεν αποτελεί την πλήρη εικόνα γιατί είναι αδύνατον να πούμε ποιος είναι καθαρά διοικητικός υπάλληλος. Η οριοθέτηση δεν είναι απόλυτη. Η διαχωριστική γραμμή δεν είναι απόλυτη, αλλά κινούμαστε μεταξύ 12 και 36% με μέσο όρο 22. Βεβαίως μπορούμε να αναρωτηθούμε γιατί συμβαίνει αυτό και να προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα. Η γραφειοκρατία αποτελεί έναν από τους λόγους. Πολλές φορές αυτό επιβάλλεται. Εγώ έχω ένα χαρτί στο γραφείο μου που έλαβα από μία εταιρεία πελάτη που δείχνει το διοικητικό φόρτο όταν θέλουμε να παραγγείλουμε έξι φλιτζάνια καφέ και τρία γεύματα για μια συνεδρίαση. Επτά ήταν τα φύλλα χαρτιού και αφορούσαν 12 υπογραφές που έπρεπε να συλλεγούν. Καταλαβαίνετε λοιπόν το επιπρόσθετο κόστος για παρόμοιες διαδικασίες για παρεμφερής διαδικασίας. Νομίζω ότι θα πρέπει να εξετάσουμε αυτή την εμβέλεια και το πεδίο εφαρμογής όπως κάνουν και όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις έτσι ώστε να μειώσουμε τη γραφειοκρατία έτσι ώστε να αποσυμφορηθεί το κόστος που μετακυλίεται στον φορολογόμενο. Πολλές φορές όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι οργανισμοί είναι ε, αρκετά μικροί και πολλές φορές απασχολούν κάτω από 50 άτομα με ένα προϋπολογισμό 20 εκατομμυρίων ευρώ. Θα πρέπει όμως να ακολουθήσουμε διαδικασία προμηθειών, προσλήψεων και ούτω καθεξής όπως αφορά τις μεγάλες ε, επιχειρήσεις και οργανισμούς. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρξει μια διαδικασία απλούστευσης και θα το προωθήσουμε αυτό στην Επιτροπή. Να υπάρξει μια διαδικασία απλοποίησης μέσα στα πλαίσια ενός ε, πλαισίου χρηματοοικονομικού κανονισμού, όπως αφορά και τον δημοσιονομικό κανονισμό. Ο κύριος Κάρλος Μοντάλβο, ο οποίος θα λάβει το λόγο, θα σας δώσει επιπρόσθετα στοιχεία για τον διοικητικό φόρτο που βλέπει ότι ισχύει στους οργανισμούς και ιδιαίτερα τους μικρούς οργανισμούς. Και ξέρω ότι υπάρχει μεγάλη καλή θέληση, πολύ καλή θέληση για να μπορέσουμε να ορίσουμε καλύτερα την πλαισίωση αυτή. Το τελευταίο θέμα αφορά τους προϋπολογισμούς των οργανισμών. Η βασική αρχή στο δημόσιο τομέα είναι πολύ απλή. Πόσο μέρος του προϋπολογισμού σας δαπανάτε και εάν είναι υψηλό το ποσοστό είναι πολύ καλό, αν όμως δεν δαπανάτε τόσο υψηλό ποσοστό γίνονται επικρίσεις. Ας πούμε ένας πατέρας δίνει 500 ευρώ στο γιο του να αγοράσει ένα ποδήλατο και ε, γυρνά στον πατέρα του και με ποδήλατο και με 100 ευρώ ρέστα. Στην κανονική ζωή θα ε, έπρεπε να συγχαρούμε το γιο. Στον δημόσιο τομέα όμως τι βλέπουμε, ότι επικρίνουμε αυτό το γιο γιατί επέστρεψε στον πατέρα με 100 ευρώ ρέστα. Δηλαδή, πώς τόλμας να γυρνάς με 100 ευρώ. Σου έδωσα τα χρήματα και έπρεπε να τα δαπανίσει. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε καλύτερους δίκτες και το ελεγκτικό συνέδριο λαμβάνει υπόψη 11 δείκτες για την διαχείριση του προπαλεγισμού και χρειαζόμαστε και ε, δείκτες απόδοσης και αποτελεσματικότητας για να δούμε πραγματικά αν υπάρχει αυτονομία του οργανισμού. Υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο σε σχέση με τους προϋπολογισμούς. Και αυτό ακολουθούν πολλές χώρες τώρα στην ε, κρίση. Οι προϋπολογισμοί των οργανισμών και άλλων επιχειρήσεων θεωρούνται ως προϋπολογισμό του παρελθόντος έτους συν κάτι και προϋπολογισμός του δύο ετών πριν συν δύο ή συν κάτι δύο φορές. Όμως, ίσως υπάρχει ρήξη των αναγκών σε σχέση με την ε, εξελικτική πορεία κάθε οργανισμού. Θα πρέπει λοιπόν να ορίσουμε εκ νέου τους προϋπολογισμούς έτσι ώστε να λάβουμε υπόψη την πραγματική εντολή Δηλαδή μιλάμε για διαδικασία μηδενικής βάσης. Δεν χρειάζεται να γίνεται κάθε χρόνο, αλλά να γίνει άπαξ διαπαντός για να ορίσουμε τις ανάγκες του εκάστοτε οργανισμού. Σε περίοδο κρίσης θα πρέπει να προβούμε σε εξοικονομήσεις χωρίς να υπάρχουν επιπτώσεις ως προς το output της, του οργανισμού αυτού, του εκάστοτε οργανισμού. Κύριε Πρόεδρε, το τελευταίο χρόνο έμαθα πολλά για τους οργανισμούς. Είναι αναγκαίοι, έχουν καλή εντολή, μπορούν ανεξάρτητα να δράσουν και να τα καταφέρουν πολύ καλά στο δημόσιο τομέα. Πιστεύω ότι τα καταφέρνουν αρκετά καλά και αποτελούν αναπόσπαστο ε, μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν συνεργαστούμε θα μπορέσουμε να ασχοληθούμε με αυτή την ιδέα του σωστού αντιτίμου για τα χρήματα που καταβάλουμε. Χαίρομαι που μπόρεσα να κάνω αυτή την εισήγηση. Δέχομαι οποιασδήποτε ερωτήσεις από τους συναδέλφους και είμαι στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστώ. Να σας ρωτήσω πότε πρόκειται να δημοσιευτούν οι εκθέσεις που οποίες μιλήσατε. Um, I cannot be absolutely... Δεν μπορώ να είμαι απόλυτα σίγουρος, ε, Πρόεδρε, αλλά πιστεύω επειδή θα αποχωρήσω από το ελεγκτικό συνέδριο το Φεβρουάριο, θα ήθελα εκείνη την περίοδο να έχουν δημοσιευθεί ή τουλάχιστον να έχει γίνει η προεργασία. Ε, ως προς τη σύγκρουση συμφερόντων έχει γίνει η εργασία, περιμένουμε και μάλλον συγγνώμη, έχει επιτελεστεί η εργασία και ως προς το benchmarking βρισκόμαστε στη στο 17ο προσχέδιο και πιστεύω ότι βρισκόμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Πιστεύω ότι το αργότερο μέχρι το ε, δεύτερο τρίμηνο του επόμενου έτους θα τα καταφέρουμε έτσι ώστε να μπορέσουμε να τα αποκριθούμε στη διαδικασία απαλλαγή του επόμενου έτους. Σας ευχαριστώ και τώρα να δώσω το λόγο στην Άννα Γιάννησεν, η οποία είναι η πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του Κοινοβουλίου για την διαθεσμική ομάδα για τις αποκεντρωμένους οργανισμούς και υπεύθυνη και από, από την Επιτροπή Προϋπολογισμού. Δέκα λεπτά έχεις, Άννα. Ευχαριστώ, Γιάν. Ε, αντικαθιστώ την Γιούτα η οποία είναι υπεύθυνη και επικεφαλής της διαθεσμικής αυτής ομάδας, η οποία είναι στο τόκο και είμαι ένα από τα πέντε μέλη που ορίστηκαν από τις διάφορες πολιτικές ομάδες. Εγώ εκπροσωπώ τους φιλελεύθερους στην διαθεσμική ομάδα εργασίας. Στην πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, ιδρύθηκε μάλλον η ομάδα αυτή, η οποία έχει την αίσθηση ότι ίσως η συμφωνία για τους οργανισμούς θα έπρεπε να επανεξεταστεί προκειμένου να συζητηθούν κάποια θέματα. Και αυτό έγινε βάσει μιας έκθεσης της Επιτροπής ΑΦΚΟ, την οποία και υπερψήφισε η Ολομέλεια, την έκθεση Παπαστάμκο, και έδωσε το πλαίσιο για αυτά που θέλαμε να συζητήσουμε. Κάποια από τα θέματα τα οποία συζητήσαμε είναι κάποια από τα θέματα τα οποία ανέφερε ο κύριος Οσί. Ξεκινήσαμε όμως λίγο πιο, σε πιο πρώιμο στάδιο από την ίδρυση των οργανισμών, γιατί ένας από τους λόγους που δημιουργήθηκε αυτή η διαθεσμική συμφωνία για τους οργανισμούς είναι ότι το Κοινοβούλιο είχε την αίσθηση ότι δημιουργούνταν όλο και πιο πολλές ε, όλο και πιο πολλοί οργανισμοί χωρίς να έχουμε επισκόπηση, χωρίς να ξέρουμε τι ακριβώς ε, γινόταν ως προς το κόστος και το όφελος, ποια θα ήταν η μεταφορά των πόρων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όλα αυτά τα στοιχεία. Άρα ξεκινήσαμε να τα συζητάμε όλα αυτά. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες οι συζητήσεις. Για παράδειγμα, η επιλογή της έδρας όπου το Κοινοβούλιο είχε την αίσθηση ότι θα μπορούσαμε αυτό να το εξετάσουμε πιο επισταμένος. Βλέπουμε ότι η έντρα επιλεγόταν ίσως όχι με κριτήρια που θα ωφελούσαν τον οργανισμό. Και θα αναρωτιόταν κανείς γιατί να μην τοποθετηθεί ο οργανισμός σε κάποιο χώρο όπου θα υπήρχε κάποια μακρά παράδοση. Για παράδειγμα, ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συντεροδρόμων στη Βαλεσιέν, στη Γαλλία. Υπάρχει κάποια παράδοση. Και αυτό ενδεχομένω να προσελκύσει και το πιο κατάλληλο προσωπικό. Ή θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι μια, ένας τέτοιος οργανισμός χρειάζεται πρόσβαση σε υποδομές, σε διεθνή αεροδρόμια, ε, ότι θα πρέπει να υπάρχουν ευρωπαϊκά σχολεία και το καθεξής. Έγιναν λοιπόν διάφορες συζητήσεις για τα θέματα αυτά. για να επιτεθούμε ίσως ε, ελαφριά, αν θέλετε, στον τρόπο που το ε, Συμβούλιο διαπραγματεύεται τις συμφωνίες αυτές, γιατί φαίνεται ότι υπάρχει μία τάση να τοποθετείται ένα οργανισμό και μετά να αφήνεται στην τύχη του διευθυντή του οργανισμού η διευθέτηση των προβλημάτων αυτών. Αντιμετωπίσαμε και άλλα προβλήματα, ωστόσο η ομάδα εργασία περιλαμβάνει και μια τεχνική ομάδα εργασία μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων, η οποία και κατήρτισε μια ολόκληρη έκθεση για τους διάφορους τομείς. Εξετάζοντας ενδεχόμενες προτάσεις για το μέλλον. Και πλέον είναι σχεδόν πλήρης και ολοκληρωμένη η έκθεση με μια περιγραφή της κατάστασης όσο έχει για τους οργανισμούς σήμερα και σχετικές προτάσεις. Επίσης, δεν συμφωνούμε απόλυτα για το πώς θα διαμορφωθεί τελικά η έκθεση θα πρέπει να το συζητήσουμε αυτό, αλλά ασφαλώς και υπάρχει επιθυμία να υπάρξει ένα μνημόνιο κατανόησης, αν θέλετε. Μια νέα διαθεσμική συμφωνία, η οποία θα προκύψει από την έκθεση αυτή και που πρέπει να σας πω ότι δίνει μια πολύ καλή επισκόπηση της κατάστασης για, τα, για τους οργανισμούς. Θα δούμε λοιπόν κατά πόσον θα καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε πριν τα τέλη του έτους. Δεν είμαι βέβαιη, αλλά αυτό παραμένει εκρεμές. Κοντεύουμε πάντως, κοντεύουμε να ολοκληρώσουμε το έργο αυτό. Να σας πω επίσης ότι συζητήσαμε το θέμα της διακυβέρνησης. για να βρούμε μια γενικότερη γραμμή για θέματα διακυβέρνησης. Υπάρχουν ασφαλώς ε, ειδικά προβλήματα σε ό,τι αφορά τα, τους οργανισμούς με τις τρεις ομάδες και τελικά καταλήγουμε να έχουμε οργανισμούς με 90 άτομα στο Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτό το εξετάσαμε ως θέμα. Το θέμα επίσης της διεύθυνσης, της διαχείρισης, το θέμα των πόρων της χρηματοδότησης συζητήσαμε. κατά πόσον θα έπρεπε να επιτραπεί στους οργανισμούς να συνεργαστούν για κάποια θέματα διευθυντικής φύσεως, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε το θέμα ότι οι οργανισμοί συχνά είναι μικροί και αντιμετωπίζουν θέματα με το προσωπικό, με τη χρηματοδότηση. Έχω επισκεφτεί και διάφορους οργανισμούς και άκουσα πάρα πολλές ιστορίες σε σχέση με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ενίοτε, που είναι ενίοτε περίεργα και ασφαλώς θα πρέπει να επιληθούν. Οι οργανισμοί λοιπόν έχουν ως σκοπό να διασφαλίσουν ότι μπορούν να ληφθούν αποφάσεις σε κοντινό επίπεδο όπως για παράδειγμα η ΕΦΣΑ, ο Οργανισμός για την Ασφάλεια των Τροφίμων, που δημιουργήθηκε μετά την ε, κρίση της υποκόντους εγκεφαλοπάθειας. Προκειμένου να μην δοθεί και πολιτική διάσταση στο θέμα, αλλά ασφαλώς υπάρχει και η πολιτική υποχρέωση λογοδοσίας. Αυτό δεν το αντιμετωπίζουμε στην έκθεση, αλλά ασφαλώς και πολλά μπορούμε να κάνουμε στο Κοινοβούλιο και ασφαλώς και στο Συμβούλιο. Ένας τρόπος αντιμετώπισης της πολιτικής λογοδοσίας είναι μέσω της διαδικασίας απαλλαγής και θεωρώ ότι αυτό αποτελεί τη βασική διαδικασία ελέγχου που διαθέτουμε στην παρούσα φάση για τους οργανισμούς. Φυσικά και οι εξειδικευμένες επιτροπές θα μπορούσαν ενίοτε να επισκέπτονται τις οργανισμούς για να ελέγχουν το έργο τους. Και ξέρω ότι κάποιες επιτροπές, όπως η Επιτροπή Περιβάλλοντος, δραστηριοποιείται ιδιαίτερα στον τομέα αυτό. Στην Ευρώπη δεν είναι δυνατόν ε, να καταγγελθεί, να κληθεί μάλλον υποχρεωτικά, όπως της είπα, ο διευθυντής ενός οργανισμού στο Κοινοβούλιο. Αλλά είμαι βέβαια ότι αν καλούσαμε τον διευθυντή ενός οργανισμού σίγουρα και θα ερχόταν. Άρα η πολιτική λογοδοσία είναι πολύ σημαντική, η πολιτική ευθύνη. Αναφέρονται στην έκθεση πολλά θέματα που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα την Επιτροπή αυτή σε ό,τι αφορά την υποχρέωση υποβολής ε, εκθέσεων. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά το προσωπικό, η κυρία Γκρέσλε ε, επέμεινε ότι για παράδειγμα θα πρέπει να ενημερωνόμαστε για τους συμβασιούχους, γιατί χρησιμοποιούνται κατά κόρον. Επίσης, ότι πρέπει να συζητήσουμε το θέμα του, της απαλλαγής. Να κοιτάξουμε τους οργανισμούς που δεν λειτουργούν μόνο με ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, με προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά αποτελούν και δημόσια σώματα. Θα πρέπει να υπάρχει κάποιος έλεγχος. Άρα, το μελλοντικό μνημόνιο συνεννόησης θα θίξει πολλά τέτοια θέματα, πολλά τέτοια προβλήματα που εντοπίσαμε για τους οργανισμούς και ξέρω ότι και το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προσθέσουν τα συμπεράσματά τους για τα αποτελέσματα, αλλά θεωρώ ότι ήταν πολύ θετικά τα αποτελέσματα και θα μας βοηθήσουν να προχωρήσουμε για να κατανοήσουμε από κοινού για το πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα των οργανισμών. Ευχαριστώ, ευχαριστώ λέει και ο Πρόεδρος. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο του Συμβουλίου. το προφέρω σωστά. Thank you very much. Dear Mr. Chairman, uh, honorable members, Mr. Um, Commissioner. Κύριε Πρόεδρε, Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο και τον εισηγητή από την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού για την πρόσκλησή σας για τη συμμετοχή αυτή. Το Συμβούλιο εκτιμά ιδιαίτερα αυτή την ευκαιρία που μας δίνεται να συζητήσουμε από κοινού τα βασικά ζητήματα που σχετίζονται με τις δραστηριότητες, το ρόλο και τη θέση των οργανισμών στο θεσμικό τοπίο της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης. Εγώ εκπροσωπώ την Προεδρία στην ε, Διαθεσμική Ομάδα Εργασίας και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε την εξέλιξη της εργασίας των αποκεντρωμένων οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, υπό την αιγίδα της διαθεσμικής ομάδας εργασίας. Μετά από την πρόσκληση του Μαΐου του 2008 από τον πρόεδρο της Επιτροπής και την διαθεσμική ομάδα εργασίας ως προς τις ε, ε, ακροάσεις ε, από τις, ε, ως προς τους οργανισμούς, αυτούς, και τη συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και Επιτροπής εξετάσαμε τα ανακύπτοντα ζητήματα ως προς την εργασία των οργανισμών αυτών. Και αυτό έγινε και μεταξύ προεδριών. Ο στόχος της συμμετοχής των εκπροσώπων του Συμβουλίου είναι να αποτιμήσουμε τη δραστηριότητα των οργανισμών με βάση μεταξύ άλλων των κριτηρίων που ορίστηκαν από το Συμβούλιο στις 17 Ιουλίου 2008 και να εξετάσουμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Κομισιόν μία προσέγγιση η οποία δεν θα είναι δεσμευτική ως προς τον ρόλο των οργανισμών αυτών. Να δούμε δηλαδή πώς δημιουργούνται πώς καταργούνται, πώς έχει η διαδικασία δημοσιονομικής διαχείρισης, την διάρθρωσή τους, τη λειτουργία και την εποπτεία τους. Στην πρώτη πολιτική συνάντηση της Διαθεσμικής Ομάδας Εργασίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή συμφώνησαν για την εκκίνηση αυτού του διαθεσμικού διαλόγου με τις, τους οργανισμούς αυτούς έτσι ώστε να δούμε κατά πόσο λειτουργούν σωστά, κατά πόσο λογοδοτούν όπως πρέπει δηλαδή κατά πόσο υπάρχει λογοδοσία και διαφάνεια των οργανισμών αυτών. Τα τρία θεσμικά όργανα αναγνώρισαν το σημαντικό ρόλο των οργανισμών αυτών στην εφαρμογή των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι ώστε να είναι ένα πιο σωστό μέσον. Μέχρι τώρα έγιναν έξι συναντήσεις σε πολιτικό επίπεδο μεταξύ Μαρτίου 2009 και Οκτωβρίου 2011. Η τελευταία συνάντηση πολιτικού επίπεδου έγινε στις 20 Οκτωβρίου 2011 υπό την Πολωνική Προεδρία. Οι συναντήσεις αυτές έχουν καθαρά τεχνικά κριτήρια και προετοιμασία. Είχαμε λοιπόν οκτώ συναντήσεις σε τεχνικό επίπεδο και η τελευταία έγινε στις 6 Οκτωβρίου. Ο συντονισμός της δραστηριότητας του Συμβουλίου έγινε με βάση, την, με, τις εργασίες, της Ομάδας Γενικών Υποθέσεων. Ασχοληθήκαμε με 34 ζητήματα, όπως συμφώνησε η διαθεσμική ομάδα. Είχαμε 34 ε, ε, δελτία και de jure αλλά και έμπρακτα μας ενδιαφέρουν λύσεις για να ορίσουμε, να προσδιορίσουμε τα προβλήματα και να βρούμε βιώσιμες λύσεις. Η εξέταση των ε, τεσσάρων τμήματων των τεχνικών δελτίων έχει λήξει. Ως προς τη διαθεσμική ομάδα βρίσκεται στο τελικό στάδιο εργασιών και τα 34 δελτία έχουν ε, εξεταστεί και η ομάδα εργασίας όρισε την κατάσταση πραγμάτων ως προς ε, διάφορες πτυχές ε, των ε, αποκεντρωμένων αυτών οργανισμών, δηλαδή διακυβέρνηση, εποπτεία και ούτω καθεξής, καθώς και μία συνεκτική εξωτερική αποτίμηση. Στο δεύτερο, σαν δεύτερο βήμα, φτάσαμε σε συνένεση ως προς τις ε, λύσεις που θα πρέπει να εφαρμοστούν για να επιλύσουμε τα οριζόμενα προβλήματα, τα προβλήματα που έχουν οριστεί. Επίσης, μας ενδιαφέρει η δημιουργία οργανισμών έτσι ώστε να δούμε ποιος είναι και ο ρόλος της χώρας υποδοχής, πώς ε, λειτουργούν τα διοικητικά συμβούλια πώς ε, έχει το έργο των διευθυντών, τα ετήσια προγράμματά τους και ε, το διοικητικό, η διοικητική υποστήριξη. Από το Σεπτέμβριο του 2011 η διαθεσμική ομάδα ασχολήθηκε με ανθρώπινους πόρους, δημοσιονομικά καθώς και ελεγκτικά ζητήματα, ζητήματα εποπτείας και ελέγχου όπως ε, βλέπετε στη τελευταία δεσμίδα δελτίων. Συζητήθηκαν τα θέματα αυτά στις 6 Οκτωβρίου και στις 20 Οκτωβρίου σε τεχνικό και πολιτικό επίπεδο. Αντιστοίχως, όπως συμφωνήθηκε στην πρώτη συνάντηση στις 10 Μαρτίου 2009, η διαθεσμική ομάδα θα πρέπει να μας δώσει συμπεράσματα μέχρι το τέλος του εγχειρήματος. Άρα, εξετάζεται το όλο θέμα και από τα τρία ε, θεσμικά όργανα με βάση την πολιτική συνάντηση που θα γίνει το Δεκέμβριο του 2011. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω και ορισμένα στοιχεία της προσέγγισης του Συμβουλίου ως προς τις αποκεντρωμένες, από τους αποκεντρωμένους οργανισμούς. Στην τέταρτη συνάντηση ε, πολιτικού επίπεδου, η Ουγγρική Προεδρία υποστήριξε ορισμένες αρχές που αποσαφηνίστηκαν σε τεχνικό επίπεδο. Καταρχήν δηλαδή, οι προτάσεις που συζητιούνται δεν αφορούν οργανισμούς που ε, ε, ασχολούνται με βάση την ΚΕΠΑ, δηλαδή το δεύτερο πυλώνα. Επίσης, ε, δεν θα εφαρμοστούν τα διάφορα στοιχεία μίας μη δεσμευτικής προσέγγισης ως προς τους προϋπάρχοντες οργανισμούς και αυτό αυτοματοποιημένα. Επίσης, οι νομοθετικού χαρακτήρα προτάσεις χρειάζονται κατά την έκβαση αυτού του εγχειρήματος, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα κάθε οργανισμού. Επίσης, δεν μπορούμε να θεωρούμε ότι υπάρχει ένα μέτρο για τα πάντα. Αυτό υπογραμμίστηκε στις συναντήσεις πολιτικού χαρακτήρα και αναγνωρίζουμε το ρόλο για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ανάγκη να είναι ένα πιο αποτελεσματικό μέσον υπ' αυτή την έννοια. Το Συμβούλιο καλωσορίζει την αγαστή συνεργασία που υπάρχει μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων στα πλαίσια της ομάδας εργασίας και ελπίζουμε ότι θα ολοκληρωθεί η εργασία το ταχύτερο δυνατόν. Επίσης, η Πολωνική Προεδρία θα αναλάβει αυτές τις εργασίες άμεσα έτσι ώστε να μπορέσουμε να οριστικοποιήσουμε αυτό το εγχείρημα πριν από τη λήξη του έτους. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ, λέει και ο Πρόεδρος. Ο κύριος Σεφκοβιτς έχει το λόγο εξ ονόματος ε, της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο Αντιπρόεδρος, για 10 λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω για αυτή την ευγενική πρόσκληση για τη σημερινή συνεδρίαση. Να ευχαριστήσω τον εισηγητή μας, τον κύριο Σταυρακάκη, για την αγαστή συνεργασία που είχαμε και να εκφράσω και την ευγνωμοσύνη μου προς τους προλαλήσαντες ε, διότι διευκόλυναν το έργο μου καθότι καλούμε να σας παρουσιάσω τις εργασίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρατηρείτε ότι υπάρχει σοβαρή σύγκληση ανάμεσα στη δική μας θεώρηση περί οργανισμών ε, για το μέλλον δηλαδή πώς ακριβώς ε, θα καταφέρουμε να επιτύχουμε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα αυτή, αυτός είναι ο στόχος ολονών. Νομίζω ότι εξετάζοντας την κατάσταση συνειδητοποιούμε πόσο σημαντικό είναι ο ρόλο των οργανισμών. Πρώτον, σε μεγάλο βαθμό συνεισφέρουν στην υλοποίηση των πολιτικών της Ένωσης και κατά αυτόν τον τρόπο βοηθούν και τους υπόλοιπους οργανισμούς καθώς και το σύνολο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να επικεντρώθει στον πυρήνα των δραστηριοτήτων, δηλαδή στην εκπόνηση των πολιτικών. Δεύτερον, προσφέρει τεχνική ε, τεχνογνωσία συγγνώμη, από εθνικό επίπεδο, περνά σε ευρωπαϊκό επίπεδο και άρα βοηθείται και η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη για το έργο τους. Ε, τρίτον, πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα, αυτό της ε, διαφάνειας, της προβολής ε, της εικόνας της Ένωσης στα διάφορα κράτη-μέλη, διότι γνωρίζετε φυσικά πως η έδρα των οργανισμών αυτών βρίσκεται ε, στα κράτη-μέλη της Ένωσης, άρα προβάλλεται το έργο τους. Ε, θα ήθελα τώρα να σχολιάσω ένα συγκεκριμένο ζήτημα σε σχέση με αυτά που ήδη ακούσαμε. Ε, η εξέλιξη των οργανισμών δεν συμβάδιζε ανέκαθεν με μια συνολική θεώρηση περί διακυβέρνησης σε επίπεδο ένωσης δηλαδή και επ' αυτού συγκλίνουμε σε σχέση με τον κύριο Όση που έχει μελετήσει με ιδιαίτερη προσοχή αυτόν τον φάκελο. Τώρα, η διαθεσμική ομάδα εργασίας ε, που συγκροτήθηκε το 2009 προσπαθεί ε, να κάνει μια δεύτερη απόπειρα, έτσι θα το έθετα. Πώς να βελτιώσει κανείς δηλαδή τη λειτουργία, την αποτελεσματικότητα των οργανισμών. Το προσπαθήσαμε το 2005, τελικά δεν τελεσφόρησαν οι προσπάθειές μας. Ε, ευελπιστούμε τώρα με αυτή τη δεύτερη απόπειρα να ε, καταλήξουμε ε, σε αυτό που θα αποκαλούσε μια κοινή προσέγγιση, μια συμφωνία, ένα μνημόνιο, πείτε το όπως θέλετε. Δηλαδή το ζητούμενο είναι να βρούμε το σωστό τίτλο για ένα έγγραφο που θα ενέχει, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, τις βασικές αρχές λειτουργίας ε, των οργανισμών, επιδιώκοντας μια αναβάθμιση αυτής της λειτουργίας όπου θα συλλέγονται επίσης ε, οι απόψεις ε, και των τριών θεσμικών οργάνων, διότι όλα τα θεσμικά όργανα έχουν σημαντικό ρόλο ε, ως προς τους οργανισμούς και το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πιστεύω πώς δοθήσεις της λιτότητας και των μέτρων περιδημοσιονομικής πειθαρχίας στα κράτη-μέλη αυτές οι προσπάθειες είναι πολύ πιο σημαντικές σε σχέση με το παρελθόν. Πιστεύουμε ότι με τις κοινέ μας προσπάθειες θα λειτουργούν πιο αποτελεσματικά οι οργανισμοί και επίσης ε, θα υπάρξει μια στενότερη συνεργασία ούτως ώστε να βελτιωθεί γενικότερα η λειτουργία και οι επιδόσεις αυτών των οργανισμών. Θα ήθελα να επιστρέψω τώρα στο έργο της Διαθεσμικής Ομάδας Εργασίας. Μετά από ιδιαίτερα εντατικές εργασίες, μετά από άοκνες προσπάθειες από πλευρά των πραγματογνωμόνων μας για τα τεχνικά ζητήματα, και μετά από την αξιόλογη ε, συνεισφορά σε πολιτικό επίπεδο στο έργο αυτή τη διαθεσμική ομάδα και εν παρόδο να ευχαριστήσω όλα τα μέλη τη καθώ και την Πολωνική Προεδρία που μετήγε σε αυτή τη συζήτηση. Όλο ιδιαίτερω ευχαριστώ την Πολωνική Προεδρία, διότι η Πολωνική Προεδρία καταφέραμε να προωθήσουμε, καταφέραμε να σημειώσουμε σημαντική πρόοδο ε, στην εξέταση του ζητήματος. Τι καταφέραμε λοιπόν να κάνουμε. Καταφέραμε να έχουμε μια γενική ανασκόπηση και μια ε, κριτική ανάλυση. Δηλαδή εντοπίσαμε ε, τα δυνατά και τα δύναμα σημεία των οργανισμών. Επίσης έχουμε στη διάθεσή μας πλέον συγκεκριμένες προτάσεις που θα μας βοηθήσουν να αναβαθμίσουμε την αποτελεσματικότητα των οργανισμών και Αυτά τα στοιχεία συνήθως συνάδουν με τις συστάσεις που είχαν ήδη καταθέσει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ελεγκτικό Συνέδριο στα πλαίσια της διαδικασία χορήγηση απαλλαγή ε, για τους οργανισμούς. Καλύπτεται πληθώρα ζητημάτων, διαχείριση των οργανισμών, παραδείγματο χάρη, τρόπο λειτουργία, έλεγχο του έργου των οργανισμών. Ε, μετά από αυτού του γενικού τίτλου, θα ήθελα να σα δώσω συγκεκριμένα παραδείγματα σχετικά με τι προτάσει και τι συστάσει που έχουμε καταθέσει. Πρώτον, η κυρία Γιάννη αναφέρθηκε ήδη σε αυτό. Νομίζω είναι ξεκάθαρο πώ ένας νέος οργανισμός θα πρέπει να θεσπιστεί μόνο μετά από αξιολόγηση αντικτύπου ε, και μετά από ε, σοβαρή ανάληψη της μελλοντικής έδρας αυτού του οργανισμού. Επίσης, ε, θα πρέπει να υπάρχει μία ρήτρα αναθεώρησης ή ρήτρα εκπνοή, sunset clause, μέσα σε κάθε πράξη συγκρότηση του οργανισμού. Τι εννοώ. Μόλις ολοκληρωθεί η εντολή του οργανισμού, πρέπει να διαπιστώσουμε αν χρειάζεται άλλη μία πενταετής περίοδο λειτουργίας, μήπως χρειάζεται τροποποίηση τη λειτουργία του οργανισμού, χρειάζεται αξιολόγηση του έργου τους, αποτίμηση του τρόπου λειτουργίας τους, γιατί μόνο έτσι θα έχουμε το ένα ικανοποιητικό επίπεδο αποτελεσματικότητας ως προς τις επιδόσεις. Μόνο έτσι θα έχουμε συνεχή έλεγχο και επιτήρηση των δραστηριοτήτων τους. Επίσης, θα έπρεπε να εξετάσουμε τη δυνατότητα συγχώνευσης κάποιων οργανισμών όταν διαπιστώνουμε ότι υπάρχει επικάλυψη ως προς τις αρμοδιότητές τους. Θα μπορούσαμε ίσως να επιτύχουμε συνεργασία ανάμεσα σε κάποιους οργανισμούς, κυρίως όταν μιλάμε για μικρού μεγέθους οργανισμούς και ο, εάν στο μέτρο που θα διαπιστώσουμε ότι με αυτή τη συγχώνευση θα ε, ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα του οργανισμού. Όπως ε, ε, είπε ο κύριος Σωσία, αξιότιμο μέλος του ελεγκτικού συνεδρίου, Μία νέα δομή διακυβέρνηση μπορεί να εισαχθεί ούτω ώστε να λειτουργούν με ομοιόμορφο τρόπο οι οργανισμοί, ε, βελτιώντα έτσι την αποτελεσματικότητά τους. Ε, φυσικά με ένα διοικητικό συμβούλιο 90 ατόμων πώς να διαχειριστεί κανείς έναν οργανισμό. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε αυτή την ε, δομή ε, των δύο στρωμάτων, δηλαδή του διοικητικού συμβουλίου και του εκτελεστικού συμβουλίου για να επιτελείται σωστά το έργο του κάθε οργανισμού. Με αυτόν τον τρόπο ε, το εκτελεστικό συμβούλιο μπορεί να εμπλακεί σε καθημερινή βάση στη διαχείριση, στα διαχειριστικά καθήκοντα που καλείται να ε, φέρει σε πέρα ο οργανισμό, παρακολουθεί εκ του σύνεγγυ τι συμβαίνει. Sometimes, uh, um... Επίσης, ε, ενίοτε επηρεάζεται αρνητικά η αποτελεσματικότητα των οργανισμών από την αλλαγή του προσωπικού μας αυτά τα διοικητικά συμβούλια των οργανισμών. Ξέρετε, ξέρουμε όλοι ότι χρειάζεται χρόνο. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να μάθουν, να καταλάβουν ε, για να μπορέσουν να είναι αποτελεσματικοί κάποια στιγμή. Νομίζουμε πως ως προς τις πολιτικές εξωτερικών σχέσεων και στις σχέσεις που έχουν εξωτερικοί οι οργανισμοί αυτοί, σε εξωτερικές Σχέσει που έχουν αυτοί οι οργανισμοί διαπιστώνουμε κάποιε δυσλειτουργίε. Δηλαδή ε, παρατηρείται μια διάσταση απόψεων, περνάει αυτό στους μα. μας, ε, ε, διότι ακούγονται απόψεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ουσιαστικά αυτό που πρέπει να επιδιώξουμε είναι να εκφραζόμαστε με μία φωνή ενώπιον των εταίρων μας. Χρειάζεται δηλαδή καλύτερη συνεργασία σε αυτό το τομέα, στις σχέσεις ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο αφενός και τους οργανισμούς αφετέρου, καλύτερο συντονισμός. Επίσης, ε, συμφωνεί η Διαθεσμική Ομάδα Εργασίας ε, πως ο ιστορικός προγραμματισμός ε, και οι γενικές προβλέψεις για τα εισοδήματα, ε, ποσοστά για τις ακυρώσεις. Όλα αυτά είναι ζητήματα που μπορούμε να βελτιώσουμε. Επίσης, ε, θα πρέπει να ε, ισχύσει μια ομοιόμορφη διαδικασία σχετικά με την υποβολή εκθέσεων. Μία ετήσια έκθεση, αυτό είναι το επιδιωκόμενο το ζητούμενο, συγγνώμη, γιατί έτσι θα βελτιώσουμε την ε, αποτελεσματικότητα των οργανισμών. Ω προ τι επιδόσει, τώρα θα πρέπει να έχουμε κάποιου βασικού δείκτε αποτελεσματικότητα. Ε, θα εγκρίνονται τα πολιετή προγράμματα και σχέση ανάμεσα στα πολιετή προγράμματα και τον προπολογισμό θα πρέπει να βελτιωθεί. Επίση, ε, θα πρέπει να βελτιώσει ο οργανισμό τη την κατάρτιση προπολογισμού βάσει δραστηριοτήτων και την υλοποίηση αυτού βάσει των δραστηριοτήτων. Πιστεύουμε πως θα πρέπει να υιοθετήσουν τώρα οι οργανισμοί αυτό το διαχειριστικό εργαλείο της κατάρτισης και υλοποίησης του προϋπολογισμού βάσει των δραστηριοτήτων. Άκουσα με ιδιαίτερη προσοχή την κυρία Γένσεν και τον συνάδελφο από την Πολωνική Προεδρία, τον κύριο Τσέρνικ, διότι Στι 20 Οκτωβρίου, τελευταίε τελευταία τη της διαθεσμικής ε, ομάδα, αποφασίσαμε να επισπεύσουμε την διαδικασία και να την ολοκληρώσουμε μέσα από αυτή την κοινή συμφωνία τη κοινέ αρχέ, ένα μνημόνιο πριν το πέρας ε, του τρέχοντο έτου. και πιστεύω ότι αυτό συνιστά σημαντικότατη πρόοδο, καμπή θα έλεγα και το συγκεκριμένο έγγραφο θα λειτουργήσει ε, και ω σημείο αναφορά για την αξιολόγηση των τωρινών οργανισμών ή κατά την εξέταση του ενδεχομένου συγκρότηση νέου οργανισμού στο μέλλον. Πιστεύω ότι σε τεχνικό επίπεδο την 1η Δεκεμβρίου θα μπορέσουμε να εργαστούμε περισσότερο εις βάθος και να βρούμε έναν τρόπο ούτως ώστε να εγκρίνουμε αυτές τις αρχές, αυτή τη δέσμη αρχών, αυτά τα συμπεράσματα σε επίπεδο διαφημιστικής ομάδας εργασίας, διότι έχουμε ήδη εργαστεί πολύ, υπάρχει σε μεγάλο βαθμό κοινή προσέγγιση και άρα θα είναι κάτι που πρέπει να αξιοποιήσουμε και να πάρει σάρκα και οστά στο μέλλον, ε, υπό αυτή τη μορφή. Πρόεδρε, κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους και πάλι από τη διαθεσμική ομάδα, από το Κοινοβούλιο, από το Συμβούλιο, την Επιτροπή και να ευχαριστήσω και τον κύριο Οσί από το Ελεγκτικό Συνέδριο για την τόσο καλή συνεργασία που είχαμε. Ο κύριος Μέλντερ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε μισή ώρα περίπου για τις ερώτα-απαντήσεις, μάλλον για τη συζήτηση. Θα ήθελε ο εισηγητής μας ε, να ε, σχολιάσει τις ε, παρεμβάσεις των εκπροσώπων των θεσμικών οργάνων πρωτού αρχή συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να καταρχήν να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους τους συμμιλητές, τους συναδέλφους που πήραν το λόγο και να διαπιστώσω για μία ακόμα φορά ότι όλοι μας αναγνωρίζουμε πράγματι τη σημασία των αποκεντρωμένων οργανισμών και ο καθένας από την πλευρά του πόσο θέλει να συμβάλλει για να, αυξήσει, να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα αυτών των κρίσιμων οργανισμών και επίσης να εκφράσω την ικανοποίησή μου ότι από όλους τους συναδέλφους αναγνωρίζεται ο ρόλος ε, των οργανισμών αυτών και ιδιαίτερα πώς μπορούν αυτοί οι οργανισμοί να βοηθήσουν ε, τις πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Thank you, Mr. Geyer, please. Ευχαριστώ, κύριε Σκάι, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χαίρομαι που σήμερα έχουμε τριγανώσει αυτή την ακρόαση γιατί είναι σωστό να εξετάσουμε και κάποια δεδομένα στη συζήτηση αυτή τα οποία συχνά ε, τα θεωρούμε αντανακλαστικά ως γεγονότα εδώ στην, ε, στο κνεβούλιο στις διαβουλεύσεις μας ε, εδώ στην Επιτροπή για το πού μπορεί να γίνουν οικονομίες διάφοροι συνάδελφοι αναφέρουν τους οργανισμούς ως απάντηση. Δεν λένε όμως ποιου οργανισμούς, τι αντίκτυπο θα έχει, σε ποια έδρα, πώς θα αλλάξει το προφίλ του, σε ποιο βαθμό θα γίνουν οι οικονομίες. Αλλά οι οργανισμοί, κατά το παρελθόν, πάντα δίναν έγκυρες απαντήσεις για το πού μπορεί να γίνουν οι οικονομίες. Χαίρομαι λοιπόν που υπησέρχονται συγκεκριμένα δεδομένα εδώ στη συζήτηση. Και που προχωράμε παραπάνω από ότι πίστευα θα προχωρήσουμε. Η έκθεση στην οποία έχω αναφερθεί σε πολλές περιστάσεις εδώ στην Επιτροπή του ελεγκτικού συνεδρίου θεωρώ ότι θα μας διευκόλυνε πάρα πολύ. Και αν σωστά κατάλαβα, ο κύριος Οσί ε, μας μίλησε για την 17η έκδοση της έκθεσης αυτής. Αυτό μας οθεί σε κάποια σκέψη. Να ρωτήσω λοιπόν τον κύριο Οσί, μα τι κάνει τόσο περίπλοκη πια αυτή την έκθεση για να έχει βγει σε 17 ξεχωριστές ε, εκδόσεις και εκδοχές. Δεύτερη ερώτηση. δεν την απευθύνω συγκεκριμένα σε κάποιον, αλλά η Αν τον Συμβούλιο, ο Αντιπρόεδρος Σεύκοβιτς ε, μας παρουσίασαν διάφορες εκτιμήσεις για το πώς έχει η κατάσταση σε αυτή τη θεσμική ομάδα εργασίας. Θεωρώ ότι συγκεντρώνουμε έτσι πολύ υλικό με το οποίο θα πρέπει να ασχοληθούμε πισταμένως. Ωστόσο, δεν κατάλαβα ακριβώς κατά πόσον το θέμα της έδρας και η κριτική για την έδρα των οργανισμών έπαιξε κάποιο ρόλο εμένα, με εκνεύρισε το γεγονός ότι η Βρετανική κυβέρνηση σε ό,τι αφορά την έδρα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων ανάγκασε να, την Ευρωπαϊκή Ένωση να αγοράσει ένα κτίριο στην πιο ακριβή πρωτεύουσα, στο Λονδίνο, για τον οργανισμό αυτό. Και είναι το κράτος μέλος αυτό, το οποίο σε κάθε ευκαιρία θέτει το θέμα των οικονομιών. Μα ποιος αποφασίζει τελικά για την έδρα και με ποια κριτήρια. Και τι περιλαμβάνεται σε μια σωστή επιλογή της έντρας. Δεν θα είχε νόημα να καταλήξουμε σε κάποια κριτήρια όπου θα πρέπει να παίζει ρόλο φυσικά για το θέμα της προσβασιμότητας αλλά και στην τελική ανάλυση της τιμής του ακινήτου. Σε ποιο επίπεδο τα πραγματευόμαστε τα θέματα αυτά στο έγγραφο εργασίας. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Η κυρία Σέσκοβα, παρακαλώ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όντως, θα ήθελα και εγώ να προσεγγίσω το θέμα αυτό από μια διαφορετική οπτική γωνία, από την οπτική γωνία του Ευρωπαίου Φορολογούμενου και από την δική μου οπτική γωνία, αν θέλετε, ως πρώην πολιτικός της τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα ήθελα επίσης να προσεγγίσω το θέμα αυτό από την πλευρά μεταφοράς αρμοδιοτήτων μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των μεμονωμένων οργανισμών. Θα ήθελα επίσης να εξετάσουμε το τι έχει γίνει στους οργανισμούς. Πάντα η δουλειά δυσκόλευε για όλους τους υπόλοιπους και ιδιαίτερα για αυτούς που ήταν στο στόχαστρο, αν θέλετε, των υπηρεσιών για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, για τους δήμους, τις κοινότητες όλους όσοι έχουν συμφέρον να προσεγγίσουν τις πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έργο λοιπόν αυτό έχει καταστεί πολύ πιο δυσχερές, πολύ πιο επαχθές. Η προώθηση της αρχικής πρόθεσης αναφέρθηκε στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μετά μεταφέρθηκε στην ιστοσελίδα του οργανισμού, μετά ε, η αρμοδιότητα αυτή πέρασε σε άλλο οργανισμό Α το κοιτάξουμε και από αυτή την οπτική γωνία. Θεωρώ ότι αυτό αποτελεί το χειρότερο μήνυμα που μπορούμε να στείλουμε προς τον έξω κόσμο, προς τους πολίτες, προς τους προλογούμενους. Είναι ό,τι χειρότερο μπορούμε να τους πούμε. Και από αυτή την πλευρά δεν μπορώ παρά να σχολιάσω τον αριθμό των οργανισμών που υπάρχουν. Κοιτάξτε, είναι και η πρώτη μου θητεία στο Κοινοβουλίο. Δεν ήμουν α, εδώ κατά τη φάση της ίδρυσης και της υπερψήπησης των οργανισμών, αλλά προσεγγίζει το θέμα και από αυτή την οπτική γωνία, αντιμετωπίζοντας το θέμα αυτό από τοπικό επίπεδο. Και μιλώ φυσικά για την ε, τσεχική δημοκρατία. Τι θα γίνει και στο μέλλον. Θα συνεχίσουν να εργάζονται οι οργανισμοί αυτοί ή μήπω θα υπάρξει και άλλη μετάθεση αρμοδιοτήτων, θα υπάρχει συγχώνευση. Η ταπεινή μου γνώμη είναι ότι οι μεμονωμένοι οργανισμοί και εμείς θα πρέπει να εξετάσουμε κατά πόσο είναι απαραίτητο να υπάρχουν μεμονωμένοι οργανισμοί ή μήπως θα έπρεπε να συγχωνευτούν με κάποιο αποτελεσματικό τρόπο. Ό,τι και να πράξουμε, Πρόεδρε, θα πρέπει να προταθεί προκειμένου όποιο επιθυμεί να κάνει αίτηση για χρηματοοικονομική υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση να ξέρει τι να κάνει. Ευχαριστώ τον Επίτροπο για την παρουσίασή του και ζητώ συγγνώμη που δεν θα ακούσω την απάντησή σας γιατί δυστυχώς ε, κάποιες επιτροπές στο Κοινοβούλιο διεξάγονται παράλληλα. Σας ευχαριστώ και τον προτέρων για την απάντησή σας. Ευχαριστώ και τώρα το λόγο έχει η κυρία Μακοβέη. <coughs> Um, you, uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω μιλήσει και στην Επιτροπή και στην Ολομέλεια σε αρκετές περιστάσεις για το θέμα αυτό. Θα είμαι σύντομη, λοιπόν. Οι πληροφορίες που έλαβε το Κοινοβούλιο από το Ελεγκτικό Συνέδριο για τους οργανισμούς και για την σχετική απαλλαγή είναι ανεπαρκέστατες για να μπορέσουμε να λάβουμε μία υπεύθυνη απόφαση ως προς την απαλλαγή. Από την απάντηση που έλαβα πριν από κάποιες ημέρες, καταλαβαίνω ότι δεν πρόκειται να λάβουμε πιο πολλά στοιχεία θα αντιμετωπίσουμε πρόβλημα και θα πρέπει να κοιτάξουμε πώς θα καταλήξουμε σε μια συμφωνία κατά την οποία θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να μας χορηγηθούν πιο πολλές πληροφορίες. Να συμφωνήσω με τους συναδέλφους σε ό,τι αφορά την έκθεση για το benchmarking για το κόστος. Δεν μπορούμε να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε το οτιδήποτε για την απαλλαγή χωρίς την έκθεση αυτή, την οποία και χρειαζόμαστε κάθε επιγόντως. Άκουσα επίσης ότι είναι η 17η έκδοση. Δεν ξέρω πόσες θα ακολουθήσουν. Επαναλαμβάνω λοιπόν το έτοιμά μου να μας χορηγηθεί η έκθεση στην παρούσα μορφή. Η δάλος θα έχει χαθεί ένα έτος σε ό,τι αφορά την απαλλαγή για τον οργανισμό. Να επιμείνω επίσης και να πω ότι δεν ήμουν εδώ εξ αρχής, αλλά συμφωνώ πλήρως με αυτά που είπε ο Επίτροπος Εύκοβιτς για το μέλλον των οργανισμών, το μέλλον των οργανισμών, ότι θα πρέπει να δούμε, να φροντίσουμε να είναι αποτελεσματικοί και αυτό να το πετύχουμε το συντομότερο δυνατόν, γιατί είναι δύσκολη η καιρή. Αντιμετωπίζουμε κρίση και οικονομική, αλλά και κρίση εμπιστοσύνη. Ο Ευρωπαίος πολίτης εμπιστεύεται όλο και λιγότερο του ευρωπαϊκού θεσμού. Κάτι λοιπόν θα πρέπει να κάνουμε, να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Έχουμε 750 εκατομμύρια συνεισφορέ ευρωπαϊκές κάθε χρόνο για τους οργανισμούς. Είναι πάρα πολλά τα χρήματα. Τι γίνεται λοιπόν με τα χρήματα αυτά. Τι θα γίνει με τα χρήματα αυτά. Όλα αυτά θα πρέπει να τα αναφέρουμε στου πολίτε. Η έκθεση δεν μου φαίνεται ότι απαντά στα θέματα αυτά. και εγώ θεωρούσα ότι αποτελούσε ένα βασικό σκοπό του εγχειρήματο. Θα σταματήσω στο σημείο αυτό και πάλι να επαναλάβω ότι ελπίζω να λάβουμε τις πληροφορίες που πραγματικά χρειαζόμαστε για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε επί του θέματος της απαλλαγής. Ευχαριστώ και τέλος. Ο κύριος Ειρενχάουζερ, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ τον Επίτροπο που έστειξε το θέμα και την, ε, το, το ενδεχόμενο της συγχώνευσης. Εγώ προσωπικά έχω καταβάλει προτάσεις για συγχώνευση και κλείσιμο μερικών οργανισμών. Να ρωτήσω συγκεκριμένα το ελεγκτικό συνέδριο ποιες, ε, ποιους οργανισμούς θεωρείτε μπορούμε να κλείσουμε συγκεκριμένα και ποιους μπορούμε να συγχωνεύσουμε και πάλι συγκεκριμένα για να έχουμε κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις. Δεύτερον, για τα κριτήρια για την έντρα. Δεν υπάρχουν επί του παρόντος. Αυτό αληθεύει και αποτελεί ένα μεγάλο πρόβλημα ότι οι οργανισμοί αλλά και οι έντρες πάντα αποτελούσαν αντικείμενο διαπραγματεύσεων στο Συμβούλιο. Ρωτώ λοιπόν συγκεκριμένα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Είναι πρόθυμο το Συμβούλιο καν να θέσει συγκεκριμένα κριτήρια για την έδρα του οργανισμού, των οργανισμών. Να μας πει το Συμβούλιο. Κατά τρίτον, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Εδώ και χρόνια είναι γνωστό το πρόβλημα αυτό και όλο κάνουμε κύκλους για το θέμα αυτό. Από το 2008 τουλάχιστον το συζητάμε. Ρωτώ λοιπόν τη συνάδελφο Γένσεν, τι συγκεκριμένες προτάσεις υπάρχουν στην ομάδα εργασίας, πότε θα τις λάβουμε. Νομίζω ότι ε, τελειώσαμε με τον κατάλογο των ομιλητών. Θα ήθελα και εγώ να προσθέσω κάτι. Ορισμένα από αυτά που θα πω ήδη προαναφέρθηκαν και ε, εγώ θεωρώ, ε, γιατί αναφερθήκατε στο Λονδίνο που είναι και η πιο ακριβή πόλη, είπατε ότι πολλές φορές υπάρχει άμεσος συσχετισμός μεταξύ έδρας του οργανισμού και της γενέτηρας και της γενέτηρας του Υπουργού Εξωτερικών, ας πούμε, της Προεδρίας ή κάποιου ηθήνοντα, υψηλόβαθμου βεβαίως. Κανένας δεν μίλησε για εκτελεστικούς οργανισμούς, executive agencies γιατί είναι εκτελεστικού χαρακτήρα και υπάρχουν ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για να επιτελέσουν ένα συγκεκριμένο ρόλο. Ο κύριος Σεύκοβιτς μίλησε για μία ρήτρα βαθμιαίας κατάργηση, sunset clause, για, τις, ε, για τους οργανισμούς εκτελεστικού χαρακτήρα. Αυτό Αναφέρθηκε αρχικά το 2004. Θα θέλαμε να ξέρουμε πόσες, πόσοι οργανισμοί εκτελεστικού χαρακτήρα υπάρχουν και πόσοι οργανισμοί θα κλείσουν τα επόμενα έτη. Ως προς αυτά που είπε η κυρία Μακοβέη, θα ήθελα το ελεγκτικό συνέδριο κάτι να μας πει ως προς το παράπονό της για έλλειψη πληροφόρησης Ίσως να την προσκαλέσετε στο Λουξεμβούργο για να σας ε, απευθύνει άμεσα τα ερωτήματα που επιθυμεί. Επίσης, πόσα προσχέδια τέλος πάντων συντάστε πριν εγκριθεί μία έκθεση. Άμεση με συγχωρείτε, λέει ο πρόεδρος. Λάθος μικρόφωνο. Θα ήθελα να δώσω το λόγο και στους άλλους ομιλητές για να απαντήσουν στα μέλη και προτείνω κάθε ομιλητής να μιλήσει για πέντε λεπτά το πολύ. Ο κύριος Οσί. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και με αυτή την ευκαιρία θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους σας, οι οποίοι υπέβαλαν ερωτήσεις. Ιδιαίτερα σκόπιμες ως προς το, την έκθεση benchmarking Νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία για την, το ελεγκτικό συνέδριο να δημοσιεύει το έργο του. Άρχισε το Μάρτιο, συλλέξαμε 6.500 μεμονωμένες πληροφορίες που έπρεπε να ελεγχθούν έτσι ώστε να γίνει η σύγκριση. Γι' αυτό και ο πολυσχηδής χαρακτήρας. Επίσης υπάρχουν 22 εταίροι όταν διενεργείται ένας έλεγχος, πολλές φορές έχουμε να κάνουμε με μία γενική διεύθυνση. Εδώ όμως είχαμε να κάνουμε με 22 συμβαλόμενα μέρη. Ο μέσος όρος για μία ειδική έκθεση από τη στιγμή της ε, έγκρισης του υπομνήματος μέχρι την εκτέλεση είναι από ε, δύο μήνες μέχρι 18. Και πολλές φορές μπορούμε να φτάσουμε και τα δύο έτη. Και όπως σας είχα πει, θέλω να μειωθεί ο χρόνος σύνταξης. Νομίζω ότι βρισκόμαστε μέσα στα χρονικά πλαίσια είχαμε 100 υποδείξεις αλλαγών εξαιτίας των ε, συμβαλωμένων μερών. Θέλουμε να τα καταφέρουμε καλά. Όπως σας σκιαγράφησα, έχουμε να κάνουμε με σημαντικά θέματα και θέλουμε να φτάσουμε σε σωστά συμπεράσματα για να έχουμε ένα υψηλό επίπεδο αποδοχής πριν, πριν δημοσιεύσουμε την εργασία μας αλλά δεν είχαμε ειδικέ εκθέσεις μέχρι πέρσι για τους οργανισμούς. Είχαμε μόνο τις οικονομικές ετήσιες εκθέσεις. Σήμερα, φέτος μάλλον, έχουμε δύο τύπους εκθέσεων για την συγκριτική αξιολόγηση κόστους, το benchmarking και δεύτερον για τη σύγκρουση συμφερόντων. Αυτές είναι εκθέσεις ειδικού και θα ήθελα στο ελεγκτικό συνέδριο να προωθήσω αυτή την εργασία. Χαίρομαι διότι υπάρχει ζήτηση της εργασίας μας και νομίζω ότι έτσι χτίζουμε ένα δυναμικό και υπήρξε υψηλή ζήτηση διότι πολύ συχνά μιλώ με τον αντιπρόεδρο, μέλη του γραφείου του, μέλη του Κοινοβουλίου και ξέρετε ότι επιτελούμε αυτή την εργασία μετά από δικά σας αιτήματα. Ελπίζω να απάντησα σε αυτό το σκέλος της ερώτησης. Κυρία Μακοβέη, θίξατε ένα θέμα σε σχέση με την απαλλαγή του 2010 και θα ήθελα να πω στους συνεδέλφους ότι δεν επήλθε αλλαγή στη προσέγγιση του ελεγκτικού συνεδρίου φέτος σε σχέση με παρελθόντα έτη. Δηλαδή, συντάσσουμε μία έκθεση τη στιγμή που έχουμε να κάνουμε με αξιόπιστα στοιχεία, τη στιγμή που έχουμε να κάνουμε με σωστά λογιστικά στοιχεία και τα ίδια στοιχεία θα δώσουμε και φέτος, όπως γίνεται διαχρονικά δεν έχει επέλθει καμία αλλαγή στις ε, πληροφορίες που ε, διαβιβάζουμε ή ε, δημοσιεύουμε. Υπάρχει μια πολύ καλή σχέση μεταξύ του εισηγητή και του μέλους του ελεγκτικού για το, τους οργανισμούς. Αυτό ισχύει με τον κύριο Σταυρακάκη και ελπίζω να ισχύει και με την κυρία Μακοβέη. Να υπάρχει εξίσου καλή συνεργασία όπως έχουμε με τον κύριο Σταυρακάκη. Μας ενδιαφέρει η απόδοση των οργανισμών ως προς τις προσλήψεις και τις δημόσιες προμήθειες. Έχει επέλθει βελτίωση διότι υπάρχει μεγαλύτερος επαγγελματισμός στους οργανισμούς γιατί εμείς μεταφερόμαστε, πηγαίνουμε επί τόπου και τους βοηθούμε με τις αποδελτιώσεις, τους λέμε ποιες είναι οι σωστές πρακτικές. Δεν είμαστε μόνο ελεγκτές, πρέπει να δώσουμε συμβουλές και βοήθεια Διαφορετικά, Πρόεδρε, απλώς ε, κάνουμε, γυρίζουμε γύρω-γύρω. Δηλαδή υπάρχει μία επανάληψη και αυτό δεν είναι καλό για το φορολογούμενο. Θα πρέπει να υπάρχουν εξελίξεις, θετικές εξελίξεις και νομίζω ότι υπήρξαν. Δεν επέκρινα έναν οργανισμό ποτέ για ε, μειωμένες δαπάνες. Ακούσατε το παράδειγμα μου με το πατέρα και το παιδί του που του δίνει χρήματα για να αγοράσει ένα ποδήλατο. Δεν θα μπορούσα να τους ε, επικρίνω κάτι τέτοιο, για κάτι τέτοιο, γιατί είμαι ένθερμος ε, καπιταλιστής, αλλά με σοσιαλιστικά ιδεώδη, λέει ο, ομιλητής. Κυρία Μακοβέη, μπορείτε να αποτανθείτε στον κύριο Σι. Συναντηθήκαμε με την κυρία Μακοβέη από τότε που ανέλαβε αυτό το ρόλο και θα ήθελα να συνεχιστεί αυτή η αγαστή συνεργασία. Μακοβέη, ευχαριστώ πρόεδρε και ευχαριστώ κύριε Οσί. Βεβαίως συναντηθήκαμε και εξετάσαμε και θέματα χρονισμού και η έκθεση συγκριτικής αξιολόγησης κόστους έπρεπε να εκδοθεί τον Οκτώβριο για να τη χρησιμοποιήσουμε για την απαλλαγή. Αυτό όμως δεν έγινε και δεν είναι σαφές γιατί. Χρειαζόμαστε όμως την έκθεση αυτή θα ήθελα να πω ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ της φετινής έκθεσης και της περσινής, γιατί πέρσι υπήρχαν επίγοντα ζητήματα προ του τους ανθρώπινους πόρους και τις δημόσιες προμήθειες. Φέτος δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Εάν λέτε ότι υπήρξε γενική βελτίωση μέσα σε ένα χρόνο, τότε θα ήθελα όλα τα μέλη της Επιτροπής αυτής να το ελέγξουν πράγματι για να δουν ότι κάτι τέτοιο ισχύει. θα έχουμε, θα έχετε πολύ, ελπίζουμε να έχετε καλή συνεργασία. Μόνο αν έχουμε την έκθεση benchmarking μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Αυτό είναι πολύ δύσκολο, αλλά μπορείτε να ζητήσετε τις πληροφορίες που θέλετε. Ευχαριστώ. Πολύ συχνά αναφέρθηκε ότι οι άνθρωποι αντιτίθενται στη δράση των οργανισμών και συμφωνώ ότι πολλές φορές ε, ε, δεν υπάρχει αρκετή γνώση για το ρόλο των οργανισμών, γιατί οι οργανισμοί περιλαμβάνουν πολλά σκέλη. Έχουμε ε, οργανισμούς δικτύωσης και δικτύων ή οργανισμούς κανονιστικού ή ρυθμιστικού χαρακτήρα. Υπάρχουν άλλοι οργανισμοί που εντάσσονται στο έργο του Συμβουλίου. Και θα θέλαμε να είναι ανεξάρτητοι αυτοί οι οργανισμοί, γιατί θέλουμε να λαμβάνουν στη, τις σωστές αποφάσεις μέσα στα πλαίσια της πολιτικής ε, λογοδοσίας. Πολλές φορές όμως δεν ε, μπορούμε να ανταποκριθούμε πλήρως, δηλαδή μπορούμε να έχουμε 27 ε, οργανισμούς τη στιγμή ε, οι οποίοι θα πρέπει να εξετάσουν αν ένα McDonald's Μακδόνελ Μπομπαρδιέ λειτουργεί καλά και είναι ασφαλές. Γιατί να το κάνουν και 27 και μην το κάνει ένας οργανισμός. Εδώ μιλάμε για επικέντρωση αρμοδιοτήτων. Γιατί πολλές φορές μπορούμε να εξοικονομήσουμε ότι όταν ε, μεταθέσουμε αρμοδιότητες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όμως γίνεται εξοικονόμηση. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη διαφάνεια και μπορώ να πω ότι στην Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού θα προσπαθήσουμε να διενεργήσουμε μία μελέτη για να δούμε κατά πόσο καρπούμεθα αυτών των ευεργετημάτων. Ως προς τα κριτήρια τώρα, για την έδρα. Θυμάμαι όταν ένας από τους οργανισμούς συστάθηκε ε, ε, σε σχέση με έναν οργανισμό ασφαλείας, τότε είπα στο Συμβούλιο γιατί στην Κρήτη, γιατί ε, στην Κρήτη και όχι κάπου αλλού. Και το Συμβούλιο μίλησε για γεωγραφική κατανομή, ότι αυτό οφειλόταν στη γεωγραφική κατανομή. Μα τότε η Ελλάδα είχε τρεις οργανισμούς και άλλες χώρες δεν είχαν. Και μου είπαν ότι δεν πρέπει να ε, αμφισβητήσω ποτέ τη σύνεση του Συμβουλίου. Οι επικεφαλής κρατών είναι οι σοφοί οι οποίοι αποφασίζουν. Αυτό μου απαντήθηκε τουλάχιστον Υπάρχει λόγο συγχωνεύσεων. Πολλοί ρώτησαν. Ναι, υπάρχει τέτοια σκοπιμότητα, αλλά δεν πρέπει να αμφισβητήσουμε τη σύνεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και πάλι, πάλι τα ίδια. Γιατί η γεωγραφική κατανομή δεν πρέπει να αντιτάσσεται στην αποδοτικότητα, αλλά όταν συζητήσαμε το θέμα των κριτηρίων, για την επιλογή έδρας. Είδαμε ότι το Συμβούλιο δεν ήθελε να επανέλθει στο ζήτημα των παλαιών οργανισμών, διότι αποτελεί μέρος ενός δούνε και λαβήν αντισταθμίσεων, αυτός πήρε το α, εκείνος το β και δεν μπορείτε να ξετυλίξετε εκ νέου το νήμα. Αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε για το παρελθόν, αλλά θα πρέπει να αμφισβητήσουμε ε, τις επίσημες αποφάσεις. Δηλαδή θα πρέπει στο δινεκές να ισχύει κάτι τέτοιο. Εγώ νομίζω ότι ορισμένες ε, ε, τριμε, ορισμένοι τριμερείς οργανισμοί θα έπρεπε να συγχωνευτούν. Σέντεφοπ, Δουβλίνο, Μπιλμπάου, ίσως θα μπορούσαν να συγχωνευτούν και να συνεδριάζουν στο Στρασβούργο. Ξέρω βέβαια ότι θα αντιταχθούν πολλά κράτη-μέλη σε αυτό. Επίσης και το Κοινοβούλιο δεν ήταν πάντα σοφό ως προς τον οργανισμό ισότητας των δύο φύλων είχαμε πει ότι δεν πρέπει να είναι έδρα η Βιέννη. Και μετά πήγε στο Βίνους. Και αυτό δεν είναι πάντα ευεργετικό τη στιγμή που υπάρχουν αυτοί οι κλειδονισμοί. Με το ελεγκτικό συνέδριο λοιπόν, με την έκθεση του ελεγκτικού θα δούμε τι γίνεται και στην διαθεσμική ομάδα εργασίας Έχουμε πολύ καλό υλικό για μελλοντική εργασία, αλλά αύριο δεν θα μπορέσουμε να παρευρεθούμε. Ευχαριστούμε. Κύριε Σέρνικ, ε, θα μπορούσατε να απαντήσετε σε ερωτήσεις. Θα μπορούσατε επίσης ε, να ρίξετε λίγο φως στην απότατη στη σοφία του Συμβουλίου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως είπε και η κυρία Γένσεν, Υπάρχουν κάποια θέματα για τα οποία δεν υπάρχει πλήρη σύγκληση απόψεων ε, στα τρία θεσμικά όργανα. Το θέμα της έδρας, μεταξύ άλλων, σε σχέση με αυτό που είπατε συνάδελφε, θα προσέθετα πως συνεχίζονται οι διαπραγματεύσει στο Συμβούλιο για να μπω και σε κάποιες λεπτομέρειες για τις θέσεις ε, των κρατών μελών στο Συμβούλιο για αυτό το ζήτημα της έδρας. Θα έλεγα ότι εμείς τουλάχιστον είμαστε σαφέστατοι και ήμασταν ανέκαθεν επανειλημμένα η Επιτροπή ακόμη και σε συνεδριάσεις πολιτικού επίπεδου ξεκαθάρισε τη θέση της. Σε πολιτικό επίπεδο λοιπόν, αλλά και σε επίπεδο διαθεσμικής ομάδας, ε, στην πολιτική συνεδρίαση που έλαβε χώρα το Μάρτιο, εμείς ξεκαθαρίσαμε ποια είναι η στάση μας. Ούτως ή άλλως το θέμα της έδρας ε, είναι μια απόφαση που ε, θα ληφθεί σε πολιτικό επίπεδο. Υπάρχει η απόφαση του 2003, να σας θυμίσω, σχετικά με την προτεραιότητα που έχουν τα νέα κράτη-μέλη για την κατανομή των εδρών υπενθυμίζω πως όλα αυτά τα ζητήματα εξετάζονται και από τα τρία θεσμικά όργανα αυτή τη στιγμή και ελπίζω ότι μετά το πέρας των διαπραγματεύσεων θα καταφέρουμε να καταλήξουμε σε μια κοινή προσέγγιση που να συνάδει και με το δίκαιο της Ένωσης. Αυτή η κοινή θέση θα συμπεριλαμβάνεται σε αυτό το έγγραφο που προαναφέραμε που θα εκπονηθεί από τη διαθεσμική αυτή ομάδα που εκπροσωπούνται τα τρία θεσμικά όργανα. Τώρα θέλω να επανέλθω σε μια παρατήρηση κυρία Σάνα Γένσεν. Κάτι που σχολιάστηκε στην αρχή της ε, συνεδρίασης. Είπατε σχολιάζοντας ε, το σχέδιο της διαθεσμικής συμφωνίας ότι ενδεχομένως δεν είναι αυτός ο στόχος μας. Εγώ θα ήθελα να τονίσω το εξής. Λόγω της ιδιαιτερότητας της δομής του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δυνάμει της εντολής των εκπροσώπων του Συμβουλίου στη διαθεσμική αυτή ομάδα που συγκροτήθηκε τον Νοέμβριο του 2008 και εγκρίθηκε φυσικά από την Κορεπέρ. Ο στόχος λοιπόν της διαθεσμικής ομάδας ε, ποιος είναι. Δεν πρόκειται καν για διαθεσμική συμφωνία. Είναι νομικά μη δεσμευτική προσέγγιση για αυτό, το ζήτημα. Νομίζω ότι χρήζει διευκρινήσεως. Αυτό δεν πρόκειται για δεσμευτικό κείμενο. Συνοψίζοντας, ε, δηλώνουμε αποφασισμένοι να καταλήξουμε σε συμφωνία, σε κοινή θέση, στο μέτρο του δυνατού, για όλο αυτό το φάσμα ζητημάτων που σχολιάστηκε. Σας ευχαριστούμε, λέει ο κύριος Μόλντερ, και ο τελευταίος λόγος στην Επιτροπή. Έχετε περίπου ένα πεντάλεπτο επίσης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα υπάρχει το ερώτημα του κυρίου Γκάγερ. Πιστεύω ότι το καλύτερο είναι να διαβάσω ε, αυτά που συμφωνήσαμε για να σας απαντήσω σχετικά με την επιλογή των εδρών για τους νέους οργανισμούς. Νομίζω ότι έχουμε συμφωνήσει ότι η απόφαση για την έδρα του κάθε οργανισμού πρέπει να λαμβάνεται πριν από το πέρασε της νομοθετικής περίοδου, ούτως ώστε να συγκροτηθεί ο οργανισμός αμελητή ε, στο χώρο της έδρας του. Ε, όχι να αποφασίζουμε εμεί στις Βρυξέλλε και να αρχίσουμε να ψάχνουμε μετά πού θα είναι η έδρα του οργανισμού. Δεύτερον, συμφωνήσαμε ότι οι αντικειμενικά κριτήρια πρέπει να συνοπολογιστούν για να επιλεχθεί η έδρα του οργανισμού, μεταξύ των οποίων έχει έγκυο ότι μπορεί να συγκροτηθεί ο οργανισμός τόπου με τη θέση σε ισχύ της πράξης ε, συγκρότησης του οργανισμού. Δεύτερον, προσβασιμότητα του χώρου. Τρίτον, κατάλληλες υποδομές για τα παιδιά του προσωπικού, διότι ανακαλύψαμε ότι κατά τη διάρκεια της ανάλυσης ανακαλύψαμε ότι μετά γίνονται αυτόχθονες εισαγωγικά οι οργανισμοί. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό. Αυξάνεται ο αριθμός των ανθρώπων από το κράτος μέλος όπου έχει την έδρα του οργανισμού, που εργάζονται στον οργανισμό, διότι είναι ευχερέστερο σε σύγκριση με συμβασιούχους ή υπαλλήλους που θα έρχονται από οποιοδήποτε σημείο της Ένωσης. Επίσης, όταν συζητείτε το θέμα της έδρες και εν ώψη της απόφασης αυτό οπωσδήποτε πρέπει να συνυπολογίζεται. Υπάρχει ένα, θα το χαρακτήριζα μάλλον πολιτικό προβληματάκι εδώ και θα ήθελα να διευκρινίσω λίγο το ζήτημα, ελπίζω να με καταλάβετε. Βλέπουμε το ισχυρό ενδιαφέρον που έχουν τα κράτη-μέλη, την αυστηρότητα που δείχνουν ως προς τους οργανισμούς και όλους τους κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία τους. Ε, και αλλάζει η στάση των κρατών μελών όταν ο οργανισμός είναι στην επικράτεια άλλου κράτους μέλους. Όταν πρόκειται για οργανισμό που λειτουργεί στην επικράτεια του ιδίου κράτους, διαφοροποιείται ξαφνικά η θέση αυτού του κράτους. Ε, νομίζω ότι αυτό που χρειάζεται είναι ε, κατανόηση, αλλοκατανόηση και κοινά κριτήρια που θα χρησιμοποιηθούν και για τους μελλοντικού οργανισμούς, αλλά όχι μόνο αυτό ε, ένα διαδικαστικό, αν θέλετε, ζήτημα στα πλαίσια της διαδικασίας αναθεώρησης της ρήτρα εκπνοής. Πώς θα γίνει η αποτίμηση της λειτουργίας του οργανισμού αν το κριτήριο της έδρας, παραδείγματος χάρη, οδηγεί σε αυξημένη ή αντίθετα μειωμένη αποτελεσματικότητα κατά την επιτέλεση των καθηκόντων του οργανισμού, όπου οπωσδήποτε θα πρέπει να συνυπολογιστεί και η έδρα στην αξιολόγηση των επιδόσεων του οργανισμού. Και νομίζω ότι οι νομοθετικές αρχές έχουν αυτή την αρμοδιότητα, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο πρέπει να ενστερνιστούν αυτήν την ε, προσέγγιση. Δηλαδή να αποφασίσουμε ποια πολιτική έμφαση θα αποδώσουμε στην αποτελεσματικότητα και την αίσια λειτουργία των οργανισμών και ε, προφανέστατα ε, κατόμοι θα φροντίσουμε ώστε να υλοποιηθεί η απόφασή μας στην πράξη. Κυρία Σέσκοβα, μας μιλήσατε για τις θέσεις του Συμβουλίου. Ο κύριος Σωσή μας έδωσε στοιχεία εύγλωτα, 47 ως 90. Γιατί διότι έχετε, ε, εκπροσωπούνται 47 μέλη, εκπροσωπείτε και, ε, ε, ε συγγνώμη, 27 κράτη-μέλη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκπροσωπούνται και τα κράτη-μέλη με κάποιους ε, εθνικούς εμπειρογνώμονες ενίοτε. Πρόκειται για διοικητικό συμβούλιο, ναι, αλλά τελικά αυτή είναι η ύπατη που θα πάρει την τελική απόφαση για τη λειτουργία του οργανισμού, για τα μελλοντικά προγράμματα που θα εγκρίνει στη λειτουργία, το έργο του οργανισμού και άρα είναι σκόπιμο να δούμε πώς αυτή η διοικητική αρχή, το διοικητικό συμβούλιο θα λειτουργεί με ομοιόμορφα για όλους τους οργανισμούς κριτήρια. Τώρα, τι περιμένουμε από αυτό το έγγραφο που θα συντάξουν από κοινού τα τρία θεσμικά όργανα στη διαθεσμική ομάδα. Ε, δεν θα είναι και επαναστατικό το κείμενο, αλλά σταδιακά ε, περιμένουμε εξελίξεις. Δηλαδή, σταδιακά θα εφαρμόζονται οι αποφάσεις ε, στους οργανισμούς, στους νέους οργανισμούς, αυτή η διαδικασία αναθεώρησης, ε, αυτή η συγκριτική αξιολόγηση θα ενταχθούν σε μια τακτική ε, αναθεώρηση της λειτουργίας των οργανισμών και πιστεύουμε πως αυτό θα ενισχύσει την κατανόηση του ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ορισμένες φορέ μέσα από συμφωνίε παροχής υπηρεσιών μπορεί να κάνει περισσότερα για τους οργανισμούς. Παραδείγματο χάρη ε, καταβολή των μισθών μέσω του PMO της αρχής ε, στο Λουξεμβούργο και τέτοια θέματα, αλλά... Όχι μόνο αυτά και η συγχώνευση μικρών οργανισμών, ε, ο προγραμματισμός των εργασιών κτλ. Δεν είναι ε, καλό να υπάρχουν οργανισμοί τόσο απομακρυσμένοι από εδώ που να μην μπορεί κανείς αυθημερών να πάει και να έρθει να επιστρέψει από τον οργανισμό. Ε, επηρεάζεται αρνητικά το έργο του οργανισμού σε σχέση με αυτό που επιθυμεί η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν είναι τόσο μεγάλη η απόσταση. Ελπίζω λοιπόν πως σταδιακά και με κάποιες προσαρμογές ε, θα ε, αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των οργανισμών. Ταυτόχρονα πρέπει να μειωθεί το διοικητικό, το γραφειοκρατικό άχθος ε, που βαρύνει τους οργανισμούς. Ας περάσω τώρα στην ερώτηση του Προέδρου. Εκτελεστικοί οργανισμοί. Ε, θέλω να τονίσω πως ε, η έκθεση και το έργο της ε, διαθεσμικής ομάδας φέρει επί των ρυθμιστικών οργανισμών και όχι των εκτελεστικών. Υπάρχει μια διαφορά, ας κάνουμε μια ιστορική αναδρομή, θα θυμάστε οι περισσότεροι ότι μιλούσαμε για μπηγόντα συστών τεκνίκ, γραφείο τεχνική αρρωγή στην αρχή. Ήταν σχεδόν ιδιωτικοί οργανισμοί που επικουρούσαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να εκτελέσει το πρόγραμμά τη και αυτό ήταν και ένα θέμα που είχε ε, ανακύψει σε σχέση με την επιτροπή του κυρίου Σαντέρ. Στο ενδιάμεσο διάστημα αναρωτηθήκαμε μήπως πρέπει να τροποποιήσουμε το σύστημα, μήπως χρειαζόμαστε μεγαλύτερη διαφάνεια και καλύτερο έλεγχο και διαχείριση για την υλοποίηση των ε, προγραμμάτων και γι' αυτό εφήβραμε και θεσπίσαμε τους εκτελεστικούς οργανισμούς. Executing μας βοηθούν να εκτελέσουμε τη μέσο συμβάσεων, ε, ε, συγγνώμη, να εκτελέσουμε το έργο που θέλουμε να κάνουμε τους το αναθέτουμε σε κάποιο συγκεκριμένο τομέα. Αυτή η ανάθεση αυτοί οι ανάδοχοι οργανισμοί βρίσκονταν πολύ κοντά ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν πολύ κοντά στον πυρήνα των ε, δραστηριοτήτων των εκτελεστικών οργανισμών. Αυτό ήθελα να εξηγήσω αυτή τη μικρή διαφορά. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εμεί ευχαριστούμε. Νομίζω για του εκτελεστικού οργανισμού θα επανέλθουμε γιατί sunset clause ρήτρα noise δεν υπάρχει για αυτού, από ό,τι κατάλαβα από αυτά που είπατε, αλλά νομίζω μεταγενέστερα θα μα απασχολήσει αυτό. Τώρα θα ήθελα να περάσω στο δεύτερο τμήμα ε, τη ε, σημερινή μα ακρόαση ε, για να μάθουμε και κάτι από τα ε, από την καθημερινή δουλειά των οργανισμών. Έχουμε ε, την καθηγήτρια Έλεν Φως από το Πανεπιστήμιο του Μάστριχτ, τον κύριο Ντανσέ από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων και τον κύριο Μοντάλβου ε, είναι ο εκτελεστικός διευθυντής της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων. Ε, έκαστος έχει στη διάθεσή του 15 λεπτά περίπου. Κυρία Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να μοιραστώ μαζί σας κάποιες σκέψεις για τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Ποια είναι τα διλήμματα και ποιες είναι οι βέλτιστες πρακτικές σήμερα, μετά από 40 χρόνια εμπειρίας με τέτοιου ε, οργανισμούς. Θα επικεντρωθώ σε πέντε θέματα τα οποία είναι αλληλοσυνδεόμενα. Το πρώτο θέμα είναι το θέμα της, του ελέγχου στους οργανισμούς ο αριθμό των μηχανισμών ελέγχου που χρησιμοποιούνται για τους οργανισμούς είναι εντυπωσιακό. Πέντε μηχανισμοί έχουν εντοπιστεί για εξάντε και ex-post έλεγχο. Έχουμε οριζόντιο έλεγχο διαθεσμικό στους οργανισμούς. Κατά δεύτερον, ξέρουμε ότι υπάρχει δικαστικός έλεγχος, ευκαιρία να καταγγελθούν ενέργειες οργανισμών που έχουν νομικό αντίκτυπο σε τρίτα μέρη. Κατά τρίτον υπάρχει διοικητικός έλεγχος για τον ρόλο των εμπλεκομένων φορέων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και υποχρέωση α, δικαιολόγησης, αιτιολόγησης. Επίσης ελέγχονται και από τον ε, διαμεσολαβητή. Επίσης έλεγχο από τα μέλη του δικτύου που έχει δημιουργηθεί από τους οργανισμούς και στα στο οποίο συμμετέχουν οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί σε αντίθεση με τους Αμερικανικούς έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν σε συνάρτηση με τους εθνικούς εταίρους. Τέλος, κάθετος έλεγχος με, μέσω του Συμβουλίου Ελέγχου και Διεύθυνσης. Υπάρχει μια σχέση δύναμης μεταξύ των οργανισμών και των κρατών μελών και μία έλλειψη υπουργικού ελέγχου στον οποίο υπόκειται συνήθως οι εθνικοί οργανισμοί. Βλέπουμε ότι υπάρχει μία, ένα μοντέλο πολλαπλών αρχών για τους οργανισμούς. Ωστόσο, ο κίνδυνος που ενέχεται είναι να υπάρχουν πάρα πολλοί υπεύθυνοι και κανείς να μην θεωρεί ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνο. Και όλοι να αποποιούνται την ευθύνη. Γι' αυτό λοιπόν θα έπρεπε να υπάρχει ένα πολυμερές σύστημα για τους οργανισμούς αυτούς. Ωστόσο, είναι απαραίτητο, αν υπάρξει ένα τέτοιο σύστημα, να κοιτάξουμε ποιες θα είναι οι αρμοδιότητες του κάθε οργανισμού. Για παράδειγμα, υπάρχει ανάγκη σαφών υποχρεώσεων για τις χρηματοοικονομικές ε, λογιστικές ε, διαστάσεις. Σε κάποιες περιπτώσεις θα πρέπει να διαπιστώσουμε ότι δεν είναι το πρόβλημα η έλλειψη ελέγχου, αλλά ο υπερβολικός έλεγχος. Για παράδειγμα, οι οργανισμοί παραπονιούνται για το υπερβολικό άχθος που έχουν επιφορτιστεί προκειμένου να πληρούν όλες τις προδιαγραφές που χρειάζεται και που έχουν τεθεί. Αυτό θα πρέπει να το αναθεωρήσουμε ριζικά. Αυτό σημαίνει επίσης ότι θα πρέπει να υπάρχουν πιο σαφείς ευθύνες για το Κοινοβούλιο σε ό,τι αφορά τον έλεγχο για τις ε, ενίοτε και εκάστοτε ενέργειες ε, των οργανισμών. Με κάποιες, ε, κάποιες επιτροπές ενημερώνονται και παρακολουθούν τις ενέργειες των οργανισμών, κάποιες άλλες όχι. Θεωρώ ότι μια καλή διαδικασία είναι η διαδικασία απαλλαγή για τα Youth in Action. Θεωρώ ότι είναι καλό το, το γεγονό ότι το Κοινοβούλιο δρά αυτόνομα. Το Συμβούλιο θα πρέπει να υποπτεύει καλύτερα του οργανισμού όταν έχει εξουσίες ορισμού και απόλυσης του διευθυντή. Επίσης, το Συμβούλιο Διευθυντών θα πρέπει να αναλαμβάνει καλύτερες ευθύνες για την καθοδήγηση του οργανισμού και θέλουμε καλύτερο ορισμό των αρμοδιοτήτων και των ευθυνών του Συμβουλίου Διευθυντών. Ποιος είναι πολιτικά υπεύθυνο το Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα μπορούσαμε να εντάξουμε τους οργανισμούς ε, στο πεδίο αρμοδιότητα της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως για παράδειγμα σε ό,τι αφορά και τα παρασυντοκτόνα. Αυτό δεν θα κάλυπτε επιστημονικές γνωμοδοτήσεις θα πρέπει να είναι πιο σαφής ο ρόλος ε, του ελεκτικού συνεδρίου σε ό,τι αφορά ε, νομικές επιπτώσεις για τρίτα, μέρα, για τρίτα μέρη. Θα ήθελα επίσης να παρατηρήσω μία τάση για άλλες μορφές ε, λογοδοσίας, την οριζόντια, δημόσια λογοδοσία που είναι απαραίτητη οριζόντιοι μηχανισμοί μέσω των οποίων οι φορείς θα μπορούν να αντιδρούν προς άλλους οργανισμούς, προς τους πελάτες τους, προς το ευρύ κοινό. Και χρειάζονται εργαλεία όπως ο κώδικας τεντολογίας, για παράδειγμα. Δεύτερο θέμα, η σχέση των οργανισμών με το κράτος μέλος όπου συστήνεται το Συμβούλιο Διευθυντών. Σήμερα αντιμετωπίζουν τρία προβλήματα το μέγεθος, τη σύνθεση και τη λειτουργία. Σε ό,τι αφορά το μέγεθος, ξέρουμε ότι σήμερα, εκτός από την ΕΦΣΑ, υπάρχουν εθνικοί εκπρόσωποι, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε κάποιες περιπτώσεις εκπρόσωποι των εμπλεκομένων φορέων και του Κοινοβουλίου. Αυτό, όπως αναφέρθηκε, οδηγεί σε συναντήσεις με 80, 90 άτομα. και στην περίπτωση αυτή δεν είναι λειτουργικά τα συμβούλια αυτά. Επιπλέον, η συχνή αλλαγή των μελών δεν συμβάλλει στη θεσμική πορεία των οργανισμών. Αυτό θα πρέπει να αλλάξει σε ό,τι αφορά τη σύνθεση τώρα. Παρατηρούμε ότι η εκπροσώπηση βασίζεται σε κριτήρια αντιπροσώπευσης, αλλά φαίνεται ότι οι εμπειρικές έρευνες έχουν δείξει προβλήματα. Δεν θα πρέπει. Θα πρέπει να κοιτάξουμε το πώς μπορούμε να εξοπλίσουμε τα συμβούλια με την εμπειρογνωμοσύνη που χρειάζεται για να εκτελέσει τα καθήκοντά της. Θα πρέπει να πούμε ότι η αντιπροσωπεύση και η εμπειρογνωμοσύνη δεν είναι πάντα αρχές που κινούνται παράλληλα. θα πρέπει να κοιτάξουμε περιπτώσεις διπλών θέσεων στα διοικητικά συμβούλια, όπου ο κόσμος απασχολείται και στο αντίστοιχο εθνικό οργανισμό. Κάποια από τα προβλήματα προφανώς ε, ανακύπτουν και στους εθνικούς οργανισμούς. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και το θέμα της έλλειψης ενδιαφέροντος προς τους οργανισμούς σε ό,τι αφορά το θέμα του μεγέθους και της σύνθεσης. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τέτοια παραδείγματα. Αλλά θεωρώ ότι θα πρέπει να εκπροσωπούνται και τα κράτη-μέλη για να ελέγχουν θέματα συμβατότητας και επικουρικότητας. Λύσεις όπως αυτή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού θα μπορούσαν να αποτελούν ένα παράδειγμα. θα πρέπει να υπάρχει η απαραίτητη δέσμευση και η εμπορογνωμοσύνη και κατά πάσα σε θέματα ηγεσία. Το τρίτο θέμα που θα ήθελα να αναφέρω δεν ε, αναφέρεται σε μια βέλτιστη πρακτική, αλλά σε μια προβληματική πρακτική σε ό,τι αφορά την, ε, το προσωπικό και την ε, διαδικασία που ακολουθείται για το ανθρώπινο δυναμικό. βλέποντας ποιο είναι ο αντίκτυπος τη σχετική πολιτική στους οργανισμούς, καταδεικνύεται ότι υπάρχει υπερβολικό έλεγχος στους οργανισμούς, γιατί η αντιγραφή ενός συστήματος σε μικρούς οργανισμούς, με λίγους ε, ε, εργαζόμενους, αναγκάζει του οργανισμούς να δουλεύουν σαν μήνυ ευρωπαϊκέ επιτροπέ. Και αυτό θα πρέπει να τροποποιηθεί. Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιλαμβάνεται το πρόβλημα που προκύπτει. Τα τελευταία δύο σημεία τα οποία θα ήθελα να συζητήσω είναι αλληλοσυνδεόμενα θέματα διαφάνειας και ανεξαρτησίας των οργανισμών. Σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επανειλημμένα αναγνωρίζει στην ομολογία ότι η διαφάνεια είναι απαραίτητη για τους πολίτες για να ελέγχουν τι ε, αρμοδιότητε της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για να ενισχύεται ο δημοκρατικό χαρακτήρα, αλλά και η εμπιστοσύνη του κοινού. Είναι προφανώς, προφανές ότι η διαφάνεια αποτελεί μια προϋπόθεση για τη λογοδοσία και τον έλεγχο. Για κάποιους οργανισμούς ε, οι πληροφορίε που διαθέτουν είναι εντυπωσιακέ. Αιτήσει, εκθέσει, αποφάσει του Διοικητικού Συμβουλίου, επιστημονικές εκθέσεις, σχέδια εκθέσεων, όλα αυτά μπορεί να βρει κανείς στο διαδίκτυο. Η διαφάνεια όμως έχει να κάνει και με τις μειονοτικές εκθέσεις, με τις ημερησίες διατάξεις και σε ό,τι αφορά και τις μελλοντικού οργανισμούς. Η αυξανόμενη διαφάνεια αποτελεί και την απάντηση στο προβληματικό σημείο της ανεξαρτησίας ε, των ε, οργανισμών που αποτελεί και το τελικό, τελευταίο μου θέμα. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η ανεξαρτησία δεν σημαίνει ότι τα άτομα δεν έχουν ε, συμφέροντα, δεν έχουν αξίες, δεν έχουν αρχές. Η ανεξαρτησία έχει να κάνει με το πώς οι επιστήμονες συλλέγουν τα στοιχεία τους ανεξάρτητα από εξωτερικές επιρροές. Και εδώ θα πρέπει να μιλήσουμε και να διακρίνουμε την ανεξαρτησία από τα βιομηχανικά συμφέροντα και τα, την ανεξαρτησία από την πολιτική. Τώρα, σε ό,τι αφορά την, ε, τα βιομηχανικά συμφέροντα, υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο είναι ευρέω γνωστό και όπω μα έδειξαν οι πρόσφατε εμπειρίε με την ΕΨΑ, εξακολουθούν να υπάρχουν τριβέ και εντάσει. Η διαφάνεια για τα μέλη, για τη δήλωση συμφερόντων των μεμονωμένων εμπειρογνωμόνων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση. Αυτό σημαίνει ότι οι οργανισμοί θα πρέπει να ορίσουν διαδικασίες για το πώς θα αντιμετωπίζουν ενδεχόμενα, ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων και θα πρέπει να, αναφέρουν και μέτρα που θα λαμβάνονται σε τέτοια περίπτωση. Για παράδειγμα, το να μην επιτρέπεται η συμμετοχή σε κάποια συνάντηση. Αυτό προφανώς ε, θα πρέπει να γίνει μετά από ιεράρχηση της σύγκρουση συμφερόντων και της δημιουργίας κάποιου πίνακα. Το προσωπικό των οργανισμών θα πρέπει να διέπεται από σαφείς ε, κανονισμούς σε ό,τι αφορά θέματα διαφάνειας, ε, συμπεριλαμβανομένων δωρεών και το καθεξής και οργανισμοί όπως η ΕΦΣΑ έχουν αρχίσει και καταρτίζουν σχετικούς κανόνες. Θα πρέπει να υπάρξει άπλατο φως λοιπόν σε όλες αυτές τις δραστηριότητε. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ λέει και ο Πρόεδρος. Και τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Τανσέτ. Thank you. Ευχαριστώ. Chairman. Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής. Χαίρομαι ιδιαίτερος που έρχομαι εδώ σήμερα για να εκπροσωπήσω τους αποκεντρωμένους οργανισμούς και ουχή τους εκτελεστικούς, όπως είπαμε, οργανισμούς. Σας ευχαριστούμε για την πρωτοβουλία. Χαίρομαι πολύ που συμμετέχω στην ε, ε, συζήτησή σας. Πιστεύω ότι το φως της δημοσιότητας ε, είναι άπλετο πλέον σε αυτά που κάνουμε, αυτά που ελέγχουμε, το πώς λειτουργούμε και άρα θα πρέπει να εντοπίσουμε τις ατέλειες να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητά μας. Δεν φοβόμαστε αυτές τις εξελίξεις, τις καλωσορίζουμε. Κυρίως σε μέρη της Ευρώπης όπου οι καιροί είναι χαλεποί, βιώνουν μεγάλες δυσκολίες οι άνθρωποι και θέλουν τα χρήματά τους να εξοδεύονται με χρηστό τρόπο και να επιτυγχάνονται οι στόχοι. Χρειάζεται λοιπόν λογοδοσία χωρίς όμως να αυξάνουμε την ε, γραφειοκρατία. Ξέρετε ότι είναι μικρού μεγέθους οι οργανισμοί, έχουν πολύ συγκεκριμένο ρόλο ακριβώς για να επικεντρώνουν τις δραστηριότητες τους ε, και να προσφέρουν τεχνογνωσία ταχύτερα και με καλύτερα αποτελέσματα. Για να το επιτύχουμε αυτό χρειάζεται άνοιγμα πνεύματος για να ε, λειτουργούμε διαλλακτικά, να εξυπηρετούμε τους πελάτες μας και διαρκώς να βελτιώνομαστε ως προς το έργο μας όλοι οι διευθυντές διευθυντές ε, των οργανισμών συμφωνούν μαζί μου. Βεβαίως, μειώνονται οι πιθανότητε επιτυχία όταν καλούμαστε να λειτουργήσουμε μέσα σε ένα γραφειοκρατικό δίκτυο. Χρειαζόμαστε στοχοθετημένα μέτρα και κάποτε μου είπε ένας διευθυντής οργανισμού ότι Χρειάζεται να υπακούσουμε σε κανονισμούς ε, που θα ίσχυαν για μια πολυεθνική εταιρεία με δεκάδες χιλιάδες εργαζομένους, όχι ένας μικρός οργανισμός με 50 άτομα προσωπικού. Επίσης, έχει αποδειχθεί ότι οι υπερβολικά περίπλοκες διαδικασίες μειώνουν την αποτελεσματικότητά μας. Ε, το ε, πιο γραφειοκρατικό είναι το ίδιο το καταστατικό Χρειαζόμαστε μέτρα που είναι προσαρμοσμένα στο μέγεθος των οργανισμών και κυρίως υπηρετούν το συμφέρον των Ευρωπαίων. Χρειάζεται έλεγχος, αλλά ταυτόχρονα χρειάζεται ευελιξία. Έτσι θα προχωρήσουμε. Ε, αυτός ε, που παίζει το βιολί αποφασίζει και ποια μουσική θα παίξει. Όμως δεν αποφασίζει το κομμάτι, ούτε τον ήχο, ε, ούτε τη χρειά που θα δώσει στο κομμάτι αυτό γιατί το λέω γιατί δεν μπορούν να λειτουργήσουν ε, ε, ελεύθερα οι οργανισμοί. Προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περαιτέρω εξορθολογισμό των αποκεντρωμένων οργανισμών τη ευρωπαϊκή Ένωση για να αυξήσει την αποτελεσματικότητά του, να του καταστήσει πιο δυναμικούς βάσει και στρατηγική Ευρώπη 2020. Συμφωνούν απολύτω οι οργανισμοί. Για να προσγειωθούμε όμω στην πραγματικότητα, προτείνουμε τρει κατευθυντηρίε γραμμέ. Πρώτον, να είμαστε υπόλογοι για τα αποτελέσματά του, το τι έχουμε επιτύχει, αλλά χρειαζόμαστε και μεγαλύτερη αυτονομία για να τα πετύχουμε αυτά. Δηλαδή, ζητούμε ένα πιο στρατηγικό ρόλο των οργανισμών. Να μην ε, εμπλέκεται τόσο πολύ η Επιτροπή στην καθημερινή διαχείριση. Δεύτερον, να είμαστε πιο αποτελεσματικοί ω προ το κόστο με απλουστευμένε διαδικασίε. Να μία ε, προσέγγιση που θα είναι προσαρμοσμένη σε κάθε οργανισμό. Τρίτον, στενή συσχέτιση ανάμεσα στο έργο που πρέπει να επιτελεστεί και στο άτομο, στα άτομα που θα επιτελέσουν αυτά τα έργα. Άρα, χρειάζεται και μεγαλύτερη διαφάνεια και εκεί επικεντρώνουμε την ενέργειά μα. Αυτέ οι τρει βασικέ αρχέ ε, συνδέονται άμεσα με τι παρεμβάσει που έχουμε ακούσει σήμερα. Βασίζονται στα αιτήματα που καταθέσαμε εμεί ε, το 2008 σχετικά με τον προγραμματισμό, την αξιολόγηση κινδύνου και τη διαχείριση των επιδόσεων. Μετά από την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου και μετά από τις συζητήσεις ε, που έγιναν στο δικαστήριο της Ένωσης. Ε, λυπάμαι, αλλά δεν αντιλαμβανόμαστε ε, πώς αυτές ε, οι συστάσεις που έχουν γίνει για τους οργανισμούς θα μας οδηγήσουν σε ένα λαμπρότερο μέλλον για να γίνουμε πιο, απο, πιο αποτελεσματικοί. Διαχείριση δύο ταχυτήτων μας προτείνεται. Αύξηση του ελέγχου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην καθημερινή εργασία των οργανισμών. Αυξημένες απαιτήσει για υποβολή εκθέσεων. Μείωση της αυτονομίας ε, των οργανισμών και μείωση των γραφειοκρατικών, των πιο γραφειοκρατικών διαδικασιών. Εμεί έχουμε συγκεκριμένε προτάσεις για βελτίωση της λειτουργίας μας και θα καταθέσουμε το τελικό μας κείμενο ε, στα τέλη του Νοεμβρίου. Χρειαζόμαστε στον πρώτο βαθμό διαβουλεύσεων, αν θέλετε, να γίνει ένας επικοδομητικός διάλογος, ώστε να καταλάβουμε με ποιο τρόπο, με ποιο μέσα θα επιτύχουμε τους στόχου που έχουμε θέσει. Οι οργανισμοί πρέπει να ασχολούνται ε, χωρί παρεμβολέ ε, με την επιτέλεση του έργου του. με το να μας δείξουν αυτά αποτελέσματα. Φυσικά θα λογοδοτούμε. Φυσικά θα μας τιμωρήσετε αν είναι ισχνές οι επιδόσεις μας. Αλλά αφήστε μας να λειτουργήσουμε. Μην ε, ε, νιώθουμε την ανάσα σας ε, πίσω μας κάθε φορά. Είμαστε οι ειδικοί και γι' αυτό και είμαστε εκεί που είμαστε. Εσείς μας βάλατε. Θα ήθελα τώρα για να είμαστε πλήρη να προσθέσουμε θέσω κάτι σε σχέση με τις πρωτοβουλίες που σας είπα νωρίτερα. Ε, το ψήφισμα το 2008, ελεγκτικό συνέδριο και δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βάσει στην έκθεση ζητήθηκε από τους οργανισμούς σε σχέση με τις επιδόσεις τους ε, συγκεκριμένα ε, μέτρα. Λοιπόν, έχουμε αναπτύξει ένα δίκτυο αποτελεσματικότητας όλων των οργανισμών για να αντιμετωπίζουμε από κοινού τις προκλήσεις και να ανταλλάσσουμε τις βέλτιστες πρακτικές. Για το συγκεκριμένο σα αίτημα χρησιμοποιούμε την κατάρτιση και την υλοποίηση του πρόγραμμα του προϋπολογισμού βάσει των δραστηριοτήτων. Ήδη εφαρμόζουμε αυτή την αρχή και ήδη έχει αυξηθεί η αποτελεσματικότητά μας. Δεύτερον, διάφοροι οργανισμοί έχουν και διαδικασία αξιολόγηση κινδύνου, ούτω ώστε τη διαδικασία αξιολόγηση να τη βασίσουν στη, στα μέτρα μετριασμού με την κέισο που ήδη ισχύουν. Τρίτον, ε, βασιζόμαστε για τις δραστηριότητες μας στο στόχο που πρέπει να επιτύχουμε και αυτό συνδέεται στενά με το λογιστικό σύστημα που χρησιμοποιούν οργανισμοί. Τέταρτον, συστήματα που βασίζονται στις επιδόσεις, ε, μετρήσιμα δηλαδή αποτελέσματα και μετρήσιμοι πόροι που χρησιμοποιούνται. Όμως, εάν διευρύνουμε αυτά τα συστήματα ώστε να αξιολογήσουμε και τον αντίκτυπο των δραστηριοτήτων των οργανισμών, τότε ανοίγουμε καινούριο κεφάλαιο. Γιατί αυτό συνιστά ένα μόνο από του παράγοντε για την αξιολόγηση του αντικτύπου του έργου των οργανισμών. Παραδείγματο χάρη σε για τη δική μου τη δουλειά θέλουμε να βελτιώσουμε το περιβάλλον και την υγεία των ανθρώπων αλλά αυτό δεν μπορεί να είναι απόρρια μόνο του δικού μας έργου ακόμη και αν συνδυαστεί το έργο του οργανισμού μα με το, τις προσπάθειες της ε, δεν πρόκειται να τα καταφέρουμε. Υπάρχουν πολλέ διαφορετικέ συνιστώσει. Εγώ και οι υπόλοιποι διευθυντές θέλουμε φυσικά να εφαρμοστούν κριτήρια αξιολόγηση επιδόσεων, αλλά θα πρέπει να επικρατήσει διαφάνεια σε σχέση με τον τρόπο αποτίμηση και αξιολόγηση ε, των επιδόσεων και θα πρέπει να συμμετάσχουμε και εμεί σε αυτή τη διαδικασία. Αν ξέρουμε ποια κριτήρια με κρίνεται, έτσι μόνο θα είμαι σίγουρο ότι σα προσφέρω αυτό που μου ζητάτε τώρα. Αν οι εκτελεστικοί διευθυντέ είναι προσωπικά υπόλογοι για την ε, απαλλαγή και για την αξιολόγηση των επιδόσεων του οργανισμού, θα πρέπει να μα δώσετε το δικαίωμα να συμφωνήσουμε κι εμεί για του στόχου που καλείται να επιτύχει ο οργανισμό και μα δώσετε και την ελευθερία, το περιθώριο ελιγμών για να επιτύχουμε αυτούς τους στόχους. Ε, η ειδική έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου για την συγκριτική αξιολόγηση ανέφερθηκε και σε ένα άλλο συγκεκριμένο σημείο που θα ήθελα να σχολιάσω. Επίπεδο δαπανών στα τέλη του έτου και μεγάλε σχετικέ μεταφορέ επιστώσεων. Ε, λοιπόν, δύο βαθμίδες, σε δύο βαθμίδε θα γίνει η αλλαγή. Πρώτον, καλύτερη διαχείριση των πόρων ε, με πιο συστηματικό τρόπο. Θα βασιζόμαστε για την κατάσταση και την υλοποίηση του προπολογισμού, όπω είπαμε, στι δραστηριότητε, activity-based. Δεύτερον, κίνητρο για του οργανισμού ε, ε, ούτω ώστε να περικόψουν τους ετησίου προϋπολογισμούς τους χρησιμοποιώντα. Ε, την επίστοση το επόμενο έτος και χωρίς να προσφεύγουν στη διαδικασία της επιχορήγησης. Για οργανισμούς όπως η δική μας με μεικτά εισοδήματα αυτό είναι ε, μια πολύ καλή λύση. Τώρα, ε, σε σχέση Σε σχέση τώρα με το τρίτο θέμα, ε, ο εξορθολογισμός, ο εξυγχρονισμός, ε, ε, για να γίνουν χοντρικά πιο δυναμικοί οι οργανισμοί, χρειαζόμαστε κατά τη γνώμη μας καλύτερο επιμερισμό ευθυνών. Ανάμεσα στα διοικητικά συμβούλια που δεν πρέπει να ονομάζονται διαχειριστικά συμβούλια, διοικητικά είναι, δεν διαχειρίζονται, διοικούν. Ε, Διαχωρισμό λοιπόν ανάμεσα στα διοικητικά συμβούλια και το, τα εκτελεστικά συμβούλια. Τα διοικητικά συμβούλια θα πρέπει να δίνουν τον τόνο, πρέπει να παίρνουν στρατηγικέ ε, αποφάσει και αυτό είναι πολύ διαφορετικό από την ε, καθημερινή διαχείριση των ζητημάτων. Χρειαζόμαστε λοιπόν αυτή την ευελιξία που σα ζητούσα προηγουμένω. Μόνο θα μπορούμε μπορέσουμε να εκτελέσουμε το καθήκον μας με πολύ πιο αποτελεσματικό τρόπο. Πρώτη θέμεθα Στι τελικέ προτάσει προ τα τρία θεσμικά όργανα μάλλον θα προτείνουμε μια ειδική διαθεσμική ομάδα εργασίας όπου θα εμπλέκονται οι οργανισμοί για να απλωστεύσουμε τους ε, το κανόνες ε, περί προσωπικού και περί καθημερινή διαχείρισης. Ελπίζω να λάβετε υπόψη αυτή την πρότασή μας. Ε, εγώ και συνάδελφοί μου φυσικά είμαστε έτοιμοι να λογοδοτήσουμε για το έργο μα αλλά μόνο αν έχουμε και περιθώριο λοιπόν, ελευθερία κινήσεων για να καταφέρουμε αυτό που μας ζητάτε. Ε, ε, ο συνάδελφος εδώ στα αριστερά που αισχάτως ε, ε, ανέλαβε εκτελεστικό ε, διευθυντή τη ΕΑΕΣ για ε, τη Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Πολυματικών Συντάξεων, κ. Μοντάλβο. Θα μα πει και εκείνο την εμπειρία του για την εφαρμογή των νέων κανόνων. Περιμένω με ελπομονησία την παρουσίασή του. Σα ευχαριστώ πάντω και πάλι για την ευκαιρία που μα δίνετε να ακουστεί η φωνή μα, οι οργανισμοί να γνωρίζετε. Είμαστε υπέρ των προσπαθειών σα για την αύξηση τη λογοδοσία και τη διαφάνεια των οργανισμών. Θέλουμε να είμαστε πιο δυναμικοί. Το κλειδί είναι να βρούμε την ισορροπία και ε, έχουμε κάθε πρόθεση να συνεργαστούμε μαζί σας για να βρούμε αυτή την ισορροπία. Ο κύριος Μόλτερ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα θα ακούσουμε τον κύριο Μοντάλβο. Ε, τώρα είναι η σειρά σας να τοποθετηθείτε. Το μικρόφωνο του μιλητή είναι σβηστό. Thank Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έλεγα ότι είναι μεγάλη χαρά και τιμή να βρίσκομαι εδώ ενώπιόν σας για να σας μιλήσω για, τη δική, για τις δικές μου εμπειρίες. Μιλάμε όμως και για κοινή ευθύνη, γιατί εμείς οι διευθυντές των ε, ευρωπαϊκών οργανισμών είμαστε και πολίτες, άρα συμμεριζόμαστε τις ε, ανησυχίες σας και θέλουμε να βελτιώσουμε τα πράγματα. Αυτό δεν σημαίνει να δούμε τις, δυσλειτουργίες. σημαίνει να δούμε τι λειτουργεί, αλλά μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα. Αυτό είναι ύψη της σημασία και θα ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας. Ποια είναι η προσέγγιση μου. Καταρχήν βασίζομαι στην πείρα μου ως Διευθυντής μη ευρωπαϊκού Οργανισμού, στη συνέχεια Ευρωπαϊκού Οργανισμού και θα σας δείξω πώς είχαν τα πράγματα πριν και πώς τώρα και ποιες είναι οι προσδοκίες μας ως Ευρωπαίοι. Δεν θέλουμε να αμφισβητήσουμε τους κανόνες, αλλά να προωθήσουμε την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα, καθώς και τη διαφάνεια και τη λογοδοσία. Πώς ε, μπορεί να γίνει αυτό. Θα, θα υποβάλω ερωτήματα που θα έθετα ως πολίτης στον διευθυντή. Πώς, τι κάνετε, πώς δαπανάτε τα χρήματά μου και πώς ξέρετε ότι αυτή είναι η σωστή λύση. Θα δείτε πώς ε, υπάρχει ε, σύνδεσμος μεταξύ αυτών των ε, ερωτημάτων. Υπάρχει δηλαδή μια αιτιώδης συνάφεια και αυτό είναι και ο λόγος υπαρξής μας. Το 2011 θέλαμε να ανταποκριθούμε στην κρίση, όπως μας όρισε η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θέλουμε να προλάβουμε και μεταγενέστερες και να μειώσουμε τις επιπτώσεις παρομοίων κρίσεων. Θέλουμε να προστατεύσουμε τους καταναλωτές, να εναρμόσουμε περισσότερο την Ευρώπη, να έχουμε περισσότερη Ευρώπη, γιατί είδαμε ότι οι σιωπηρές ή οι απομονωμένες απαντήσεις δεν επιλύουν το πρόβλημα και θέλουμε να υπάρχει και χρηματοοικονομική σταθερότητα. Αυτός είναι ο ρόλος μου, η αποστολή μου και εδώ γίνεται η πραγματογνωμοσύνη. Και αυτό είναι και το προφίλ αυτό που θέλω να προσλάβω. Γιατί μέσω του οργανισμού θα δώσω προσθέμενη αξία στους πολίτες και θα κάνω τη διαφορά. Και γι' αυτό θα υπάρχει αυτός ο οργανισμός. Πώς ε, δαπανούμε τα χρήματα του Ευρωπαίου πολίτη. Υπάρχει το θέμα των προμηθειών, του ελέγχου, των δαπανών και του δημοσιονομικού ελέγχου. Ας αρχίσουμε με τα δημοσιονομικά, με το προϋπολογισμό. Θεωρώ ότι ξεχνάμε τι σημαίνει προϋπολογισμός. Ο προϋπολογισμός δεν είναι παρά ένα δημοσιονομικό μέσο για να παράγουμε το πρόγραμμά μας, να εκτελέσουμε το πρόγραμμά μας και έχει σημασία το περιεχόμενο και η διαδικασία. Αν δείτε τη διαδικασία και σας ενδιαφέρει η έγκριση, θα πρέπει να έχετε ένα πρόγραμμα εργασίας με βάση τις ανάγκες και έτσι θα μπορέσετε να κατανείμετε τα χρήματα. Ποια ήταν η πρώην κατάσταση και ποια η νυν. Πριν είχα ένα πρόγραμμα εργασίας, ένα προσχέδιο και βλέπαμε τι πόρους έχουμε στη διάθεσή μας για να προβούμε σε μία ευθυγράμμιση. Τώρα έχουμε μια διαφορετική κατάσταση, όπως στις 15 Φεβρουαρίου κάθε έτους πρέπει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει ένα προσχέδιο προϋπολογισμού για το επόμενο έτος, το οποίο σημαίνει σήμερα στις 21 Νοεμβρίου ήδη εργάζομαι για τον προϋπολογισμό μου του 2013. Εργάζομαι στον ε, οικονομικό τομέα ε, εν μέσω κρίσης και δεν ξέρω τι θα κάνω τον επόμενο βήμα, τον επόμενο μήνα, με συγχωρείτε. Είναι πολύ νωρίς να πούμε οτιδήποτε, γιατί ο προϋπολογισμός μου εντάσσεται στη Γενική Διεύθυνση Αγοράς και μέχρι το Φεβρουάριο θέλουν να ξέρουν κατά πόσο ε, συνάδει με τις ανάγκες. Η πρώτη πρόταση προϋπολογισμού δεν προέρχεται από εμένα, αλλά από τη μελέτη αντικτύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αν το σκεφτείτε λοιπόν και δείτε ποιος είναι ο τελικός στόχος του προϋπολογισμού, βλέπουμε ότι υπάρχει αντιστροφή του βασικού κύκλου ως προς την ανάπτυξη και την αποδοτικότητα. Ποσά τώρα. Χρειαζόμαστε επαρκή ποσά, αλλά πόσα χρήματα. Ο κύριος Οσί μίλησε για τους δείκτες δαπανών. Αν το δούμε αυτό σαν μέτρο ε, αποτελεσματικότητας μπορεί να είναι αντιπαραγωγικό. Το τέλος του έτους θα έχω ένα αριθμό εκτέλησης και θα έχω ένα αποθεματικό του 20% του μελλοντικού προϋπολογισμού. Όλα τα άλλα θα αποδοθούν στα μέλη. Πώς έχει η κατάσταση εάν ο δείκτης δαπανών δεν είναι αρκετά καλός, δεν θα μου δώσει απαλλαγή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα μου ασκηθεί πίεση να μειωθεί ο μελλοντικός μου προϋπολογισμός. Ας δούμε ένα παράδειγμα. Είναι ο πρώτος μου χρόνος και δεν θα μπορώ να έχω υψηλό δίκτυ εκτέλεσης στον ε, τομέα του κεφαλαίου 3. Γιατί? Γιατί μιλάμε για ένα φιλόδοξο πρόγραμμα, το οποίο θα πρέπει να εκτελέσω με βάση την εργασία μου και τις ε, προμήθειες και τις αναθέσεις. Εάν δούμε λοιπόν την ε, λήψη αποφάσεων και μετά την ανάθεση, είναι αδύνατο να ανταποκριθώ. Άρα θα προσπαθήσω να αλλάξω το σύστημα έτσι ώστε να έχω επαρκή δίκτυ δαπανών ή να είμαι υπεύθυνο και να πω ότι για να δαπανίσουμε τα χρήματα θα πρέπει να γνωρίσουμε το πλέον αποδοτικό τρόπο δαπάνης. Είπα ότι υπάρχουν λάθος κίνητρα πολλές φορές. Την προηγούμενη εβδομάδα στην Επιτροπή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μίλησα, μιλούσα για δίκτυ εκτέλεσης και τους είπα πόσοι γνωρίζετε ότι για το 2012 το δεύτερο χρόνο που υπάρχουμε εμείς μου προτείνεται μία μείωση του προϋπολογισμού. Και θα ήθελα να σας εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου γιατί είπατε ότι αυτό δεν είναι αποδεκτό στον, στον οργανισμό μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Είναι πολύ καλό παράδειγμα. Ένα άλλο παράδειγμα όταν μιλάμε για τον προϋπολογισμό θα πρέπει να δούμε το προσωπικό. Θα πρέπει να έχουμε την περιγραφή τη θέσης, της θέσης και να ξέρουμε γιατί προσλαμβάνεται κάποιος. Πέρσι όταν συμμετείχα σε μία μη κερδοσκοπική επιχείρηση είχα την ίδια προσέγγιση, αλλά αν εξαιτία της κρίσης ένα από τα θεσμικά όργανα μου ζητούσε να κάνω κάτι διαφορετικό, από το να προσλάβω κάποιον ε, ε, άλλον έκανα έναν ανασχηματισμό αρμοδιοτήτων και ενέτασα ναι, στοιχεία σε χαρτοφυλάκια ακόμα και όταν δεν είχαν προσληφθεί γι' αυτό. Αυτό θα πει αποδοτικότητα. Άρα θα πρέπει να έχουμε ευελιξία. Θα πρέπει να μιλάμε και για έλεγχο και εποπτεία, γιατί έχει σχέση με την λογοδοσία. Όλοι πιστεύουμε στη λογοδοσία και τον έλεγχο. Από τότε που εργάζομαι στον οργανισμό Ξέρετε ποια αρχή εκφράζω, την αρχή των τεσσάρων ανθρώπων. Δηλαδή, ε, εγώ ή ο αναπληρωτής μου, α, τι κάνουμε, τι κάνουμε, αναθέτουμε. Τώρα όμως χρειαζόμαστε τέσσερα άτομα. Είναι αποδοτικό. Όχι, λέω, ας αρχίσουμε με τέσσερις και επειδή θέλω να έχω μεγαλύτερη αποδοτικότητα, θα προβάλλω μια πρόταση για να πω κατά πόσο θα πρέπει να είναι τέσσερις. Γιατί όχι μόνο έχουμε την ε, αρχή ενός συστήματος του ΑΒΑΚ και θα πρέπει να έχουμε και την αρχή των υπογραφών επί χάρτου. Έχει νόημα. Αυτό ακριβώς κάνουμε και θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τη μεγαλύτερη κρίση που γνωρίσαμε μέχρι τούδε. Μερικοί μιλάνε για μεγαλύτερη κρίση από αυτή του 29. Ξέρετε ποιες ήταν οι τρεις πρώτες μου προσλήψεις στον οργανισμό μου. Ένας εμπειρογνώμονας, ένας αναλογιστής, ένας που θα ήξερε την πραγματικότητα των χρηματοοικονομικών οργανισμών. Όχι, ήταν ένας λογιστής, ένας υπεύθυνος για τα χρηματοοικονομικά και ένας υπεύθυνο αναθέσεων. Και πιστεύω στους ελέγχους. Έχουμε το ελεγκτικό συνέδριο, έχουμε τον εσωτερικό έλεγχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχουμε την Όλαφ, τον Ομπούτσμαν ε, και έχουμε μία επιτροπή ελέγχου, ποιοτικού ελέγχου, για να πούμε πού μπορούμε να βελτιώσουμε τα πράγματα και εκεί που λειτουργούν και εκεί που δεν λειτουργούν καλά. Επίσης θέλουμε τα μέλη μας που καταβάλουν το 60% των εισφορών να δουν αποτελεσματικότητα, όπως θέλετε και εσείς σαν Κοινοβούλιο, σαν Ελεγκτικό Συνέδριο και σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα δεν αμφισβητούμε τους κανόνες, τους ακολουθούμε και τους αναθεωρούμε. Μπορούμε να αλλάξουμε τη σχέση κόστους-οφελίας. Εάν ναι, τότε θα προβάλλουμε μία πρόταση έτσι ώστε να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Πώς δαπανώνται τα χρήματα, ανάθεση. Η ανάθεση έχει σχέση με τη διαφάνεια. Προσωπικά μπορώ να σας πω ότι ήμουνα καθηγητής ε, συμβατικού και εταιρικού δικαίου, αλλά πάντα υπάρχουν όρια. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ευελιξία. Υπάρχουν τα κατόφλια και υπάρχουν και τα κίνητρα. Ας αρχίζουμε με τα κίνητρα. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τη χρηματοοικονομική κρίση. Άρα χρειάζομαι πληροφορίες, θα πρέπει να προσλάβω που μπορεί να γίνει είτε με το Bloomberg είτε με Thomson Reuters. Υπάρχουν ε, συγκεκριμένοι κανόνες ανάθεσης. Πάω στο Bloomberg και τους λέω ε, κερδίσατε πρέπει να ακολουθήσετε αυτούς τους όρους. Εγώ λέω όχι. Θα ακολουθήσετε τους δικούς μου κανόνες. Τι κάνω εγώ, αμφισβητώ το σύστημα και λέω ότι θα ακολουθήσω τους κανόνες του Bloomberg ή δεν θα λάβω τις πληροφορίες. Χρειάζεται θάρρος. Και εγώ είπα ναι, εφόσον χρειάζομαι αυτές τις πληροφορίες για να κάνω τη δουλειά μου, θα αναλάβω έναν κίνδυνο είναι σωστό κίνητρο. Όχι. Τα κατόφλια. Ποια κατόφλια πρέπει να διανύμεται και να επαναδιανύμεται. Πολλές φορές χρειάζονται αναθέσεις και επιμέρους αναθέσεις. Θεωρείτε ότι ο πάροχός σας ε, θα τα καταφέρει και καθυστερεί δύο μήνες. Τι μπορείτε να κάνετε σε αυτή την περίπτωση παρόχων, μπορείτε να αναθεωρήσετε ή βρισκόσαστε σε μία στάση αναμονής. Μάλλον θα πρέπει να κάνετε το δεύτερο. Ένα άλλο θέμα που θα ήθελα να δω είναι οι δαπάνες. Μιλάμε για αναγκαίες και μη αναγκαίες ε, δαπάνες. Ε, αυτές που μπορούμε να αποφύγουμε και αυτές όχι. Γιατί ακόμα και σε ποσά που δεν είναι σημαντικά θα πρέπει να έχετε υπόψη αυτή τη διάκριση για να τα καταφέρνετε. Ποια είναι μια δαπάνη που μπορεί να αποφευχθεί. Επειδή λειτουργεί σωστά το σύστημα για να μετατρέψουμε τα γερμανικά ε, συμβόλαια σε ευρωπαϊκά χρειάστηκε να καθυστερήσω κατά μία εβδομάδα για την διαδικασία διοδότησης από τις Βρυξέλλες και γι' αυτό έπρεπε να πληρώσω την κοινωνική πρόνοια αυτού του, του προσωπικού γιατί δεν θα ήταν ε, προστατευμένη. Είναι κάτι το αναγκαίο ή όχι. Δεν το ξέρω. Ας δούμε τι κάνουμε στον παρόντα οργανισμό. Μιλάμε για κατάρτιση από τους ευρωπαϊκούς ε, οργανισμούς. Μου λένε ας πούμε ότι μπορεί η κατάρτιση κρατάει ένα μήνα, αλλά καταβάλλεται ολόκληρο το χρόνο. Όχι, τότε θα περιμένω τον επόμενο χρόνο. Γιατί στο παρελθόν πήγαινα στην ΕΚΤ και ζητούσα από τη Φραγκφούρτη να γίνει ένα swap μεταξύ της ε, κατάρτισης που υπήρχε και αυτής που προσέφερα, έτσι ώστε να δούμε κατά πόσο μπορεί να γίνει ανάθεση ή όχι. Αυτές είναι οι καταστάσεις που αντιμετωπίσαμε και αντιμετωπίζουμε και δεν θέλω να επικρίνω το σύστημα. Θέλω να επικρίνω τον ε, τρόπο λειτουργίας, δηλαδή πώς μπορούμε να δεχτούμε το γενικό πλαίσιο όταν φτάνουμε στις λεπτομέρειες. Το τελευταίο ζήτημα, πόσο γνωρίζω ότι βρίσκομαι στο οδό. Οι πολίτες το ξέρουν. Πρέπει να υπάρχει πλήρης διαφάνεια και λογοδοσία. Είμαστε υπέρ, αλλά είμαστε και υπέρ της ευελιξίας στην πλαισίωση, διότι οι κανόνες σημαίνουν χρήμα, στοιχίζουν και μπορείτε να πείτε πολλές φορές εντάξει αξίζει ας δαπανίσουμε ή μπορείτε να πείτε υπάρχει άλλος τρόπος για να φτάσουμε σε, αυτό το, σε αυτή την έκβαση. Άρα δεν ισχύει ένα μέτρο για όλα γιατί διαφορετικά δεν είμαστε αποδοτικοί και αυτό δεν είναι καλό για τους πολίτες. Και με βάση αυτά που είπε ο Επίτροπος θα ήθελα όλοι να είμαστε φιλόδοξοι έτσι ώστε να μην είμαστε μεγάλοι επαναστάτες. Να πάρουμε, να κάνουμε τα μικρά βήματα που στο τέλος κάνουν τη διαφορά. Γι' αυτό θεωρώ ότι πρέπει να βρίσκομαι ενώπιόν σας και να καταστήσουμε τα πράγματα καλύτερα. Thank you very much. Then we have... Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και έχουμε ακόμα μισή ώρα έρωτα Και θα ήθελα να δώσω το λόγο... Α, όχι, δεν θέλει ο συγκεκριτής το λόγο. Θέλει κανεί άλλο ένα άλλο βουλευτής, να θέσει ερώτηση στους τρεις ομιλητές. Μα μου δίνετε το λόγο, ευχαριστώ πολύ. Συχνά ακούω πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση και πόσο ε, επαχθείς είναι οι κανόνες. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω ποιου κανόνε να αλλάξουμε, γιατί είμαι και εισηγήτρια σε θέματα προπολογισμού και δέκα φορέ έχω θέσει την ερώτηση αυτή σε διαφορετικά άτομα, σε διαφορετικέ χρονικέ στιγμέ. Θα ήθελα αυτό το γενικό παράπονο να το συγκεκριμενοποιήσουμε με συγκεκριμένε απαντήσει και σε ό,τι αφορά τον κανονισμό του προσωπικού. Θα ήθελα να με διαφωτίσετε στο τι μπορούμε να βελτιώσουμε. Ευχαριστώ. Μάλιστα, κυρία Μακοβέλη. Σας ευχαριστώ πολύ. Να ρωτήσω την κυρία Φως κάτι συγκεκριμένο. Αναφέρθηκε σε θέματα διαφάνειας. Ανέφερε ότι σε κάποιους οργανισμούς είναι πολύ καλά η διαφάνεια. Μπορείτε να μας πείτε σε ποιους οργανισμούς δεν υπάρχει διαφάνεια. Και επίσης, Μία δεύτερη ερώτηση. Δεν υπάρχουν παραδείγματα οργανισμών με καλές ή κακές πρακτικές. Μόνο ακούμε κάποιες γενικές εκτιμήσεις, κάποια γενική αξιολόγηση. Δεν μπορούμε έτσι όμως να εργαστούμε, γιατί σε κάποιους οργανισμούς υπάρχουν προβλήματα, σε κάποιους άλλους υπάρχουν άλλα προβλήματα. Μα να κατανομάσουμε συγκεκριμένα τους οργανισμούς. Και τέλος ένα σχόλιο. Στο μέλλον Ίσως να πρέπει να καλέσουμε πιο πολλούς αξιόλογους, ε, πιο, συγγνώμη, ανεξάρτητους ε, εμπειρογνώμονες ε, για να κάνουν αξιολόγηση της κατάστασης, γιατί μόνο η κυρία Τεφός είναι εξωτερική. Θα ήθελα ίσως στην επόμενη ακρόαση να καλέσουμε πιο πολλά άτομα εξωτερικά. Ευχαριστώ. Ο κύριος Όντι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. όχι από όταν ε, πρωτοεκλέγινα, ε, αλλά τέλος πάντων εδώ και καιρό έχω εμπλακεί ενεργά στη ζωή αυτών των οργανισμών και ειλικρινά με τη σημερινή ακρόαση επιβεβαιώνονται οι επιφυλάξει και οι ενδιασμοί μου. Ε, κοστίζουν ακριβά οι οργανισμοί, 30% διοικητικά έξοδα με την πάροδο των ετών δεν διαπιστώνουμε στην ουσία αν υπάρχει προστιθέμενη αξία. Μας είπαν ότι λειτουργούν αυτοί οι οργανισμοί σαν μικροεπιτροπές. Δύσκολα μπορεί να το διαπιστώσει κανείς. Από τα διοικητικά συμβούλια απουσιάζει χαρακτηριστικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όχι, δεν ισχυρίζομαι ότι θα πρέπει να εκπροσωπείτε το Κοινοβούλιο. Θα μπορούσατε να μας προσκαλέσετε με την ιδιότητα του παρατηρητή για να δούμε Έχουμε την αίσθηση εμεί ότι λειτουργούν ως ε, ε, μικρές ε, διακρατικές μικροδομές αυτοί οι οργανισμοί. Δηλαδή η επικοινωνία με το Κοινοβούλιο χωλαίνει. Χρειαζόμαστε περισσότερα στοιχεία για να διαπιστώσουμε αν υπάρχει προστιθέμενη αξία με αυτόν τον πολλαπλασιασμό αυτών των μικροδομών και βλέποντα ε, τις τίτλους ε, των 20 τόσων οργανισμών συν του εκτελεστικού οργανισμού για την έρευνα. Βλέπουμε Εκτελεστικό οργανισμό για την καινοτομία και την έρευνα. Εκτελεστικό Οργανισμό για την έρευνα. Εκτελεστικό οργανισμό ε, για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνα σίγουρα σε κάτι χρησιμεύουν αυτοί οι τρεις οργανισμοί, αλλά τι καταλαβαίνουν οι πολίτες από αυτά, τίποτα. Για την υγεία. Ευρωπαϊκός οργανισμός για την Υγεία στο χώρο εργασία. Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Πρόληψη και τον Έλεγχο των Νόσων. Ευρωπαϊκός οργανισμός Φαρμάκων. Ευρωπαϊκός οργανισμός για την Επισητιστική για την Ασφάλεια των Τροφίμων. Εκτελεστικός οργανισμός για την Υγεία. Πέντε, έτσι, ήδη. Ε, ε τώρα, εκτελεστικό οργανισμό για για την ε, κατάρτιση έχουμε ευρωπαϊκό οργανισμό. Τώρα δεν είναι οργανισμός, είναι ευρωπαϊκό κέντρο για την επαγγελματική κατάρτιση. Για τις αξίες, ε, ε, οργανισμός για τις θεμελιώδεις αξίες Ευρωπαϊκής Ένωσης και προσθέσαμε και ένα Ινστιτούτο για την ισότητα των δύο φύλων. Μα η ισότητα δεν είναι θεμελιώδες δικαίωμα. Εγώ ήμουν εισηγητής για την αξιολόγηση του 7ου ερευνητικού πλαισίου της Ένωσης. Οι εμπειρογνώμονες που έκαναν την αξιολόγηση ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σταματήσει με αυτέ τι μικροδομές ε, διότι έχουμε την εντύπωση ότι δεν υπάρχει πιλότο πια μέσα στο αεροπλάνο ε, οι Αμερικανοί θέλουν να μάθουν ποιο είναι το αφεντικό εν πάση περιπτώσει στην Ένωση δεν ξέρουμε που μα πάνε τα τέσσερα εγώ έρχομαι από ένα κράτο μέλο όπου πραγματικά η λογική μα είναι αυτή τη ε, κεντρικής ε, δεν λέω ότι χρειάζονται αφεντικά για όλα αλλά προσοχή ας μην αντιταχθούμε σε αυτή την ιδέα, διότι επιδιώκουμε την αποτελεσματικότητα και οι πολίτες πρέπει να καταλάβουν ότι χρησιμοποιούνται σωστά ε, τα χρήματά τους και χρειαζόμαστε ευρωπαϊκούς οργανισμούς και όχι διακρατικούς. Κυρία Κρέσλη, θα σας δώσουμε το λόγο, αλλά ο κ. Γκάιρ έχει ζητήσει πρώτος. Αν παρακολούθησα σωστά τις διαπραγματεύσεις, το κόστος, το 30% είναι ε, μάλλον η πιο φιλόδοξη, πιο υψηλός αριθμός που έχω ακούσει. Εγώ άκουσα ένα 12%. Δεν ξέρω αν είναι υπερβολικά αισιόδοξα αυτά. Συμφωνώ απόλυτα. Στο σημείο αυτό να γίνουν κάποιες ε, διαχωρισμοί. Αλλά θα πρέπει να ε, θέσουμε και σαφώς τις αρμοδιότητες από πλευράς της Επιτροπής μας και όταν μου δίνεται η αίσθηση ότι διαβάζω μία αναφορά για μία, ένα, αν θέλετε, μία ανταλλαγή στο Συμβούλιο θεωρώ ότι η ευθύνη για την ε, αναποτελεσματικότητα δεν βρίσκεται εδώ στην Επιτροπή μας, αλλά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Διαβάσα την ε, απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ποια θα πρέπει να είναι ε, το συμπέρασμα για την μη χορήγηση απαλλαγής τη ΣΥΠΟΛ. Τι να σας πω, ούτε εγώ ξέρω. Δεν προβλέπεται από τις συνθήκες. Σκεπτόμενος ότι θα έχουμε συζητήσει τα θέματα αυτά στην Επιτροπή μας και ότι έχουμε ασκήσει σαφή κριτική, θα πρέπει να πω ότι η ΣΕΠΟΛ δεν είναι και πιο μεγάλος οργανισμός και δεν εκπροσωπείται, ε, δεν εκπροσωπούνται και τα 27 κράτη-μέλη. θα συμμετέχει ίσω και η γερμανική αστυνομία, όλα είναι πολύ σωστά, αλλά ποιο έχει τελικά τον χρηματοοικονομικό έλεγχο, την χρηματοοικονομική εποπτεία για τον οργανισμό αυτό. Άρα ανακύπτει το θέμα του πού έγκαιται η ευθύνη. Ρωτώ λοιπόν την κυρία Φως, τι θα μας συστήνατε ως εξωτερική ως προς την πολιτική προσέγγιση για να ξεκινήσει μια συζήτηση σε ό,τι αφορά τις ευθύνες ελέγχου και εποπτείας από τη πλευρά θεσμική. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κυρία Κρέσλερ, πάλι. Ο συναδέλφος Οντί μας μίλησε για το θέμα αυτό. Κατά πόσο οι κοινέ πρωτοβουλίες τεχνολογίας έχουν συμπεριληφθεί δημιουργήθηκαν πέντε νέα σώματα στα οποία χορηγούμε απαλλαγή και ανησυχώ ιδιαίτερα <coughs> μετά από αυτά που είπε ο συνάδελφος ότι, ότι τα έργα αυτά θα διωγγώνονται και θα πηγαίνουν. Εγώ προσωπικά ανησυχώ γι' αυτό, δεν ξέρω. Το ομολογώ. Μάλιστα, λέει ο πρόεδρος, δεν βλέπω κανείς άλλος. Α, η κυρία Γιάνσεν. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξή, αν μου επιτρέπετε. Χάρηκα που άκουσα και τις τρεις εισηγήσεις. Νομίζω ότι ήταν ιδιαίτερα ωφέλιμες. Αλλά ο τελευταίος ο μιλητής, ο οποίος έχει πολύ ενδιαφέρουσες εμπειρίες και θα πρέπει να σας πω ότι κάποιες εξ αυτών τις έχω ακούσει ήδη και στο παρελθόν. Ένας οργανισμός που έπρεπε να προκηρύξει διαγωνισμό για 30 κινητά τηλέφωνα και δεν ήταν πολλές οι εταιρείε εκείνες οι οποίες θέλησαν να συμμετάσχουν και οι υπάλληλοι χρησιμοποιούσαν αναγκαστικά τα δικά τους τηλέφωνα για να λειτουργήσει το οργανισμό. Τέτοια προβλήματα ανακύπτουν συνέχεια. Αλλά να ρωτήσω σε ό,τι αφορά τον κανονισμό για το προσωπικό και για τις προσλήψεις. Πώς λειτουργεί και σε ό,τι αφορά τη χημική βιομηχανία, γιατί υποτίθεται ότι απασχολείται εμπειρογνώμονες, τους καλύτερους επιστήμονες στον τομέα της χημικής βιομηχανίας στην Ευρώπη, άτομα ειδικά και εμπειρογνώμονες και σε οικονομικά ζητήματα. Λειτουργεί τελικά ο κανονισμό αυτός, μπορείτε να προσλάβετε αυτούς που χρειάζεστε. Μάλιστα, λέει ο Πρόεδρος. Δεν βλέπω κανέναν άλλον. Να, θέλει το λόγο. Άρα θα καλέσω τους τρεις ε, ομιλητές να απαντήσουν και μετά θα δώσω το λόγο στον Επίτροπο για να απαντήσει στον κύριο Γκάιερ και στον κύριο Γκρέσλα και στον κύριο Ντί. Έχετε το λόγο, κυρία Φως. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ για τις ερωτήσεις που μου θέσατε. Σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια, δεν είπα πραγματικά ότι η διαφάνεια είναι σε πολύ καλό επίπεδο σήμερα. Απλά ήθελα να πω ότι κάποια, κάποιοι οργανισμοί έχουν σπουδαίες ιστοσελίδες και δίνουν πολλές πληροφορίες στους πολίτες. Δεν μπορώ να σας αναφέρω τώρα ποιες, ε, ποιοι οργανισμοί δεν είναι διαφανείς. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι πρέπον. Δεν ξέρω, αυτό απαντάει το ερώτημά σας. τώρα, σε ό,τι αφορά τα μαθήματα που μπορούμε να αντλήσουμε εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να εστιαστούμε στην πολιτική ευθύνη και στην πολιτική λογοδοσία και ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου, αλλά να βρούμε και άλλε μορφέ λογοδοσία. Και αυτό θεωρώ ότι αποτελεί ένα βασικό μήνυμα, ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι ε, οριζόντιας ε, λογοδοσίας, οριζόντιων ευθυνών, όπου θα μπορούσε, για παράδειγμα, να υπάρχει λογοδοσία προς τους άλλους οργανισμούς, προς τους πελάτες, προς το κοινό, σε ό,τι αφορά τώρα το όλο σύστημα λογοδοσίας και το γεγονός ότι δεν υπάρχει ένα βασικό σύστημα οργανισμών και υπουργική ευθύνη για τους οργανισμούς στην Ευρώπη. Νομίζω ότι και η βιβλιογραφία διχάζεται στο σημείο αυτό. Το καλύτερο μοντέλο το οποίο καλύπτει την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το μοντέλο πολλαπλής αρχής. Ότι υπάρχουν διάφορα θεσμικά όργανα τα οποία είναι υπεύθυνα για τους οργανισμούς και ότι αυτό θα πρέπει να το σεβαστούμε γιατί ανήκει στον ίδιο το χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά αν σεβαστούμε την παράδοση αυτή θα πρέπει να καταστήσουμε σαφέστερες και τις αρμοδιότητες, τις ευθύνες, το τι έχει ανατεθεί σε κάθε θεσμικό όργανο ως ευθύνη. Ο κ. Στανσέ. Να επανέλθω στο θέμα αυτό για την ερώτηση της ε, διαφάνειας και της σύγκρουσης των συμφερόντων, γιατί οργανισμός μου είναι ένας από τους τέσσερις οργανισμούς που έχει εξεταστεί από το ελεγκτικό συνέδριο για τέτοια θέματα και να θυμάστε ότι είμαστε σχετικά καινούριο οργανισμός, 4,5 χρόνια έχουμε. Και η πρώτη πολιτική ήταν ένα θέμα, μια πολιτική που σχετιζόταν με θέμα σύγκρουση συμφερόντων. Ισχύουν κάποιοι κανόνες, αλλά προφανώς και μπορεί να υπάρξει βελτίωση. Το να γνωρίζουμε αυτό και έχουμε βελτιώσει και τις σχετικές δηλώσεις. Έχουμε συστήσει μια ανταλλογική επιτροπή για ενδεχόμενες ανησυχίες. Έχουμε καταρτήσει ένα κώδικα διοντολογίας. Έχουμε θέσει κανόνες για περίπτωση σύγκρουση συμφερόντων και αντιμετώπιση τους ε, με επαγγελματικό τρόπο, καταβάλουμε τέτοιες προσπάθειες για να προληφθεί τέτοια περίσταση, τέτοιο πρόβλημα, ώστε να δεν έχει εμφανιστεί τίποτε. Παρ' όλα αυτά είναι χρονοβόρα η διαδικασία. Σε ό,τι αφορά την επιθυμία να κατονομαστούν συγκεκριμένα οι οργανισμοί που τα πάνε άσχημα, Νομίζω ότι ως κοινοβούλιο θα πρέπει να αποφύγετε να παίξετε το παιχνίδι του τύπου, γιατί ο τύπος ενδιαφέρεται μόνο για τις ε, κακές ειδήσει. Δεν αναφέρει τίποτα για τις ε, εύρυθμα λειτουργούσες ε, υπηρεσίες. Ενδιαφέρεται μόνο για οργανισμούς όπου παρουσιάζονται προβλήματα, όπου κάποιος παραβίασε τους κανόνες. Άρα θα ήθελα να εντοπίζετε τα μεν, αλλά παράλληλα να αναγνωρίζετε και το καλό έργο που γίνεται στους οργανισμούς, για στην τελική ανάλυση αυτός είναι ο σκοπός μας. Σε ό,τι αφορά την απλούστευση των κανόνων. Πρότεινα να καταρτιστούν προτάσεις για το πώς μπορεί να απλοποιηθεί η κατάσταση για μικρότερους οργανισμούς. Υπάρχουν εκατοντάδες κανόνες τους οποίους μπορούμε να εξετάσουμε προκειμένου να βρούμε τρόπο απλούστευσης και σε ό,τι αφορά τον οικονομικό κανονισμό. Αναφέρθηκαν διάφορα παραδείγματα. Δεν θα μπορούσαμε τώρα φυσικά να παριθμίσουμε όλες τις δυνατότητες, αλλά καλό θα ήταν τα τρία θεσμικά όργανα να κάτσουν στο τραπέζι διαπραγματεύσεων με τους οργανισμούς και να κάνουν προτάσεις απλούστευσης προκειμένου να γλιτώσουν πολύ επιπλέον κόστος. Νομίζω ότι αυτό θα ήταν πολύ θετικό για την πρόσληψη. Έχω... Ήμουν υπεύθυνο για την πρόσληψη 500 ατόμων στη Φιλανδία, 2.000 χιλιόμετρα από τις Βρυξέλλες. Ε, νομίζω ότι προσελκύσαμε αρκετό κόσμο. Το πρόβλημα είναι πόσο μακρά είναι η διαδικασία, γιατί παίρνει πάρα πολύ χρόνο μέχρι ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίε αυτέ και υπάρχουν καθυστερήσει. Κάτι άλλο που είναι πάρα πολύ σημαντικό και ήθελα να το αναφέρω, η απέτηση τρίτης γλώσσας για τις Είναι δύσκολο γιατί οι επιστήμονες μας, οι εμπειρογνώμονες μας δουλεύουν στα αγγλικά και προτού πάρουν πραγωγή πρέπει να, πάρουν, να μιλούν μια τρίτη γλώσσα και δεν βλέπουν οποιαδήποτε ανάγκη να μάθουν μια τρίτη γλώσσα και αυτό συχνά τους αποθεί. Αυτό είναι διαφορετικό. Σε ότι, δεν ισχύει μάλλον σε ό,τι αφορά το διοικητικό προσωπικό, τους ε, αυτή μάλιστα, όπως και στην Επιτροπή, να μιλούν τρεις γλώσσε. Αλλά όταν μιλάμε για κορυφαίους επιστήμονες, όταν προαπαιτούμε μια τέτοια γλώσσα, πολύ απλά χάνουμε πολλούς επιστήμονες. Και αυτό είναι το τίμημα του να ζητάμε έναν ομοιόμορφο κανόνα για όλους, που να ισχύει για όλους. Ο κύριος Μοντάλβο, ευχαριστώ. Να απαντήσω σε αυτό που με ρώτησε η κυρία Καταρχάς, να πω το εξή. Είπατε ότι το έχω ακούσει και στο παρελθόν. Ναι, ελπίζω σε τέσσερα χρόνια να μπορούμε να είμαστε σε θέση να το θέσουμε το θέμα αυτό. Γιατί σε σύγκριση με το γάμο μου, ε, τι να σα πω, εγώ θεωρώ ότι υπάρχει πρόβλημα σαν γάμο όταν δεν τίθενται τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Φυσικά υπάρχουν θέματα τα οποία μπορούν να βελτιωθούν. Αλλά δεν θα ήταν πολύ πιο απλό να έρθω και να σα διαβάσω πέντε λεπτά κάτι μια ομιλία την οποία μπορεί και να μην καταλαβαίνω καλά-καλά. Θα ήταν πιο εύκολο από το να κάνω μια σύγκριση με το πώς ήταν η ζωή πριν και πώς η ζωή ήταν μετά. Για το θέμα των προσλήψεων, τη συγκεκριμένη ερώτηση που μου θέσατε. Τρία θέματα θα ήθελα να θίξω. Καταρχάς, ε, στην θέματα πρόσληψη. Ο οικονομικός κλάδος απαιτεί εμπειρογνώμονες. Στο δικό μου τομέα κοστίζει μια περιουσία. Ο αναλογιστής, για παράδειγμα, κοστίζει πάρα πολλά χρήματα. Ξέρετε ότι ε, εργαζόμαστε βάσει ενός σχεδίου με διάφορες θέσεις, το οποίο καταρτίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μας το προτείνει και στην αρχή έχουμε πολλούς βασικούς εμπειρογνώμονες, έτσι είναι η ορολογία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουμε και διάφορους εμπειρογνώμονες, δύο ερωτήσει. Καταρχάς, από πλευρά ε, διαστητική. Ποιο θεωρείται ότι θα είναι πιο δύσκολο να προσλάβω ένα AD10, AD11 ε, ε, όχι έναν ND5. Έχω δυσκολίε σε ό,τι αφορά του κορυφαίου εμπειρογνώμονε, γιατί δεν υπάρχει ισορροπία μεταξύ αυτού που ζητάω και αυτού που προσφέρω. Δεν έχω πρόβλημα όμω να προσλάβω του πιο νέου. Χρειάζομαι όμω και του δύο. Χρειάζομαι μια ισορροπία. Κατά δεύτερον, μετά από την σύσταση του σχεδίου ίδρυσης υπάρχει ένας κανόνας που δεν με αφήνει να προσλάβω πάνω από 20% του συνολικού προσωπικού ως βασικούς εμπειρογνώμονες. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό και πολύ λογικό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε, μία, σε έναν οργανισμό που δημιουργήθηκε το 2011, το 2014 να μπορώ να προσλάβω μόνο ε, 20% άτομα με κορυφαία εμπειρία, η κατάσταση είναι πολύ μακριά από το να είναι ιδανική. Και όπως σας είπα, ότι έρχομαι εδώ απλά για να σας παρουσιάσω τα προβλήματα και να βρούμε λύσεις. Γι' αυτό σας παρακαλώ, βοηθήστε μας. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, και πριν δώσω το λόγο στον Επίτροπο, θα ήθελα το Συμβούλιο μήπως να απαντήσει. Όχι το ελεκτικό συνέδριο. Μάλιστα. Um, just to say that... Ήθελα μόνο να πω πως ε, οι απόψεις που εκφράστηκαν σήμερα εδώ ταυτίζονται με τις απόψεις που ακούω όταν επισκέπτομαι εδώ και χρόνια τους οργανισμούς κάθε εβδομάδα. Ο κύριος Μοντάλβο και ο κύριος Ντάσετε είπαν πράγματα γνωστά. Οι οργανισμοί και το ελεγκτικό συνέδριο δεν νομίζω να έχουν άπειρε δυνατότητε. Ε, έχουν άπειρε δυνατότητε αλλαγή ε, και μπορούν να εξοικονομήσουν χρήματα και να γίνουν πιο αποτελεσματικοί. Πρόεδρο. Ελπίζουμε η μέθοδος δειγματοληψία να είναι εξίσου καλή όσο η δική σας. Θα ακολουθήσουμε, ξέρετε, τις συστάσεις σα για βελτίωση τη λειτουργία των οργανισμών. Ο κύριο Εύκοβιτ, τώρα ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις διάφορες απόψεις, προσεγγίσεις ε, που εκθέσατε εδώ. Ο κύριος Οσί είπε νωρίτερα και ήθελα να το επαναλάβω Εξάλλου το ακούσαμε και από τους ε, εκτελεστικούς ε, διευθυντές. Είπε λοιπόν ότι όλα αυτά είναι γνωστά και επαναλαμβάνονται. Δηλαδή κάθε οργανισμός ε, ισχυρίζεται, επικαλείται την ιδιαιτερότητά του για να δικαιολογήσει μια ειδική μεταχείριση. Άρα πρέπει να έχουμε ειδικέ μεταχειρήσει για όλους αυτούς τους οργανισμούς αν ακολουθήσουμε τη λογική. Ναι, μεν, αλλά θα πρέπει να τηρούμε για τους κανόνες που ισχύουν για όλους. Ε, γιατί για τον απλό λόγο ότι μας χρηματοδοτούν τα δημόσια κονδύλια. Άρα ε, ε, ε κρατικές προμήθειες, διαγωνισμοί, ελεγκτές και ούτω καθεξής. Φυσικά στον ιδιωτικό τομέα είναι πιο ευέλικτα τα πράγματα. Δεν είμαστε όμως ιδιωτικό τομέα, ακόμη και εκεί συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Θα πρέπει λοιπόν να διαπιστώσουμε με ποιο τρόπο μπορούμε να τηρήσουμε αυτούς τους κανόνες περί ελέγχου, εποπτείας, χρηστής ε, οικονομικής διαχείρισης, ενώ ταυτόχρονα ε, θα δώσουμε μία απάντηση ε, σε αυτά τα προσκόμματα που υπάρχουν και μας απομακρύνουν από την υψηλότερη αποτελεσματικότητα και καλύτερες επιδόσεις των οργανισμών. Ταυτόχρονα δεν πρέπει να αποχωρήσουμε με την αίσθηση ότι δεν εκτιμά κανείς το έργο των οργανισμών. Δεν ισχύει αυτό. Φυσικά χρειαζόμαστε του οργανισμού και νομίζω όλοι το αναγνωρίζουν αυτό, την τεχνογνωσία του. χρειαζόμαστε την ε, ανεξάρτητη γνωμοδότησή του, χρειαζόμαστε αυτά που κάνουν και χρειαζόμαστε και περισσότερα μάλιστα. Ε, θέλουμε μια αυξημένη αποτελεσματικότητα, αυξημένε επιδόσει και αυτό είναι και το θέμα μα. Πώ μπορούμε να βελτιώσουμε του όρου εργασία των οργανισμών, με ποιο τρόπο μπορούμε να βελτιώσουμε τι συνθήκε λειτουργία του ε, για να αναμείνουμε και ε, καλύτερα αποτελέσματα μια πιο αποτελεσματική έκβαση στις εργασίες ε, που επιτελούν. Εδώθη μεγάλη σημασία στην προετοιμασία αυτού του τελικού εγγράφου των τριών θεσμικών οργάνων. Ε, πού, σε ποιο σημείο έχουμε φτάσει, πού ε, παρατηρείται πρόβλημα, συμφόρηση, τι μπορούμε να κάνουμε, ούτως ώστε να βελτιωθεί η συνεργασία ανάμεσα στην Επιτροπή ε, και τους οργανισμούς. Πρώτον, About uh, training, recruitment. Uh, πρώτον, σε σχέση με τη στελέχωση βάσει της διαδικασίας ε, προκήρυξης διαγωνισμού για κρατικές προμήθειες σήμερα. Έχουμε τις οδηγίες ε, για την παροχή υπηρεσιών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, όταν διαπραγματευόμαστε ε, από απόφαση πλαίσιο, ούτως ή άλλως εντάσσουμε τους οργανισμούς σε αυτές τις αποφάσεις βάσει του κανονισμού περικρατικών προμηθειών λόγω των προβλημάτων που έχουν εντοπίσει οι διευθυντέ ω προ τον ετήσιο προγραμματισμό. Και άρα επιλέξαμε ε, τα πολυετή προγράμματα. Πιστεύουμε ότι πρέπει να έχουν στρατηγική θεώρηση των πραγμάτων ε, οι οργανισμοί. για να μπορέσουμε, νομίζω, αν επιδιώκουμε να έχουμε ένα στρατηγικό χαρακτήρα προγραμματισμό σε επίπεδο ένωση, α αρχίσουμε από του οργανισμού. Ε, έτσι θα επιτύχουμε καλύτερο προγραμματισμό. Για τη στελέχωση αυτών των οργανισμών. Νομίζω ότι θα πρέπει να συνεργαστούμε με το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αρχής γενομένου στο Δεκέμβριο και σίγουρα το επόμενο εξάμεινο και κατά πάσα πιθανότητα το επόμενο έτος. Το επίπεδο ε, των μισθών. Πώς θα έχουμε τους ευέλικτου δυνατούς υποψηφίους και πώ ε, θα πληρώσουμε αυτούς τους μισθούς. Εντάξει, όλοι θέλουν τον καλύτερο. Πώς Ε, θα πληρώσει για όλα αυτά. θα πρέπει να δούμε πώς θα χειριστούμε αυτή την οικονομική διάσταση της ε, πολιτικής τελέχωσης των οργανισμών. Να εξετάσουμε το ενδεχόμενο ε, εκπαίδευσης, παραδείγματο χαρή. Ε, πρόσκληση εμπειρογνώμων, όπως κάνουμε και στην Επιτροπή. Αν ήταν η Επιτροπή να προσλαμβάνει όλους τους εμπειρογνώμονες από... Ε, καταλαβαίνετε... Φυσικά υπάρχει ότι δεν γίνεται. Υπάρχει η ευελιξία του 20% για τους οργανισμούς, δηλαδή μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι ε, απουσιάζει πλήρως η ευελιξία. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε τους όρους εργασίας και συνεργασίας με τους οργανισμούς. Κάνουμε μια πρόταση για περαιτέρω απλουστεύσεις. Έγιναν πολλές αναφορές στους κανόνες της Επιτροπής, στο ε, κανονισμό προσωπικού για τους μεγάλους οργανισμούς κτλ. Εμείς προτείνουμε, ε, ε, ε των αναλογιών να εφαρμόζονται ε, αυτοί οι κανονισμοί. Δηλαδή να βρίσκουμε τρο, προσπαθούμε να βρούμε τρόπους για να βελτιώσουμε το σύστημα. Τέλος πάντων τώρα κάτι που μου ήρθε για τα πειθαρχικά συμβούλια παραδείγματος χάρη ή οποιαδήποτε άλλα συμβούλια. Μπορούμε να ε, θεσπίσουμε κοινά τέτοια συμβούλια. Και αν ε, το καλοσκεφτούμε, θα βρούμε και άλλες τέτοιες δραστηριότητες που θα μπορούσαμε να ε, εκτελέσουμε από κοινού στο μέλλον. ε, αν δείτε τις προτάσεις μας για τον ε, κανονισμό προσωπικού, θα, δούμε, θα δείτε ότι προτείνουμε μια νέα κατηγορία προσωρινών υπαλλήλων συμβασιούχων για τους οργανισμούς θα έχουν καλύτερε ε, πρόπτικες για την επαγγελματική του σταδιοδρομία, έτσι θα γίνεται πιο εύκολα η απόσπαση σε άλλους οργανισμούς και άρα θα ενισχυθεί η σταθερότητα του σε επίπεδο προσωπικού, θα ε, αυξήσουμε τα θέλγητρα ε, για τους υποψηφίους. Νομίζω ότι θα καλωσορίσει το προσωπικό αυτές τις προτάσεις γιατί πρόκειται για καταγγελίες που συχνά έχουν καταθέσει. Τα τελευταία δύο χρόνια καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να αναλύσουμε την κατάσταση, να υποβάλουμε τι καλύτερε δυνατέ προτάσει και ελπίζουμε στο μέλλον με λίγη καλή ή πολύ καλή πολιτική βούληση και καλύτερη διαθεσμική ε, συνεργασία, καλύτερη συνεργασία ανάμεσα στου οργανισμού και την Επιτροπή, θα έχουμε μια πληρέστερη εικόνα, σαφέστερη εικόνα για να αξιοποιήσουμε και να θέσουμε σε εφαρμογή τα πορίσματα αυτή τη ε, έκθεση τη διαθεσμική ομάδα. Πρόεδρος, ε, ο εισηγητής μας ε, θα ήθελε τον ε, λόγο για να κάνει κάποια καταληκτικά σχόλια. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, αν θα έπαιρνα τον λόγο πριν από τον Επίτροπο, μάλλον το υποθετηθώ διαφορετικά. Με όσα είπε ο Επίτροπος, ο αντιπρόεδρο τη Επιτροπής, στα περισσότερα σημεία με βρίσκουν σύμφωνο και επομένω δεν νομίζω ότι θα πρέπει να τα επαναλάβω. Η σημερινή συζήτηση πάντως αποδείχθηκε ότι ήταν μια πολύ χρήσιμη συζήτηση και είναι πολύ παρήγορο και πολύ θετικό ότι τρεις διαφορετικοί θεσμοί με τους, ε, με τα, με τους οργανισμούς βρίσκονται σε απόλυτη συνεργασία, ανταλλάσσουν απόψεις με βασικό στόχο την σύγκληση των απόψεων και την αύξηση της αποτελεσματικότητας πάντοτε με κριτήρια διαφάνειας και λογοδοσίας Πιστεύω και με αυτό θα τελειώσω, είμαι όπως προανέφερα απόλυτα στη γραμμή του κυρίου Επιτρόπου ότι ναι μεν υπάρχουν διαφορετικοί οργανισμοί ε, σε διαφορετικές θέσεις, ε, με διαφορετικό, τρόπο, με διαφορετικό αριθμό διοικητικών συμβουλίων, με πάρα πολλά προβλήματα. Θα πρέπει όμως να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε να γίνει μια ομογενοποίηση, να γίνει μια εναρμόνιση ε, των κριτηρίων τα οποία θα μπορούν να εφαρμοστούν ε, αν όχι σε, όλα, ε, σε, αν όχι σε όλους τους περισσότερους οργανισμούς. Ευχαριστώ και πάλι τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής, τον κύριο Όση από το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο, το Συμβούλιο, τη συνάδελφο κυρία Γένσεν, τους αγαπητούς συναδέλφους για την, και πολύ ενδιαφέρουσες ε, ερωτήσεις και απόψεις που κατέθεσαν και φυσικά τους ε, εκλεκτούς καλεσμένους μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. I, we have come at the end of... Σας ευχαριστούμε και φτάσαμε και στο τέλος αυτής της τόσο ενδιαφέρουσας ε, ακρόασης. Όταν ήμουν εισηγητής για τον προπολογισμό το 2004, το έτος της διεύρυνσης δηλαδή, ο προπολογισμό για το διοικητικό κόστο τη Επιτροπής αυξήθηκε κατά 0,8% λόγω της διεύρυνσης και ο προπολογισμό των οργανισμών κατά 4,3% διότι έπρεπε να έχουν διερμηνία κτλ. όλοι οι οργανισμοί. Πρέπει να δούμε λοιπόν αν αξίζει η επένδυση σε σχέση με το αποτέλεσμα για τους εκτελεστικούς οργανισμούς. Τώρα επίσης το 2004 καταλήξαμε σε διαθεσμική συμφωνία και σαφέστατα είπαμε ότι ε, οι εκτελεστικοί οργανισμοί είναι περατοί, ε, ε, δηλαδή διαρκούν 6-7 χρόνια μέχρι να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα. Αλλά παρόλα αυτά εξακολουθούν να υπαρχουν εξαιρετικά εκτελεστικοί οργανισμοί και άρα χρειάζεται έρευνα επ' αυτού. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ε, συμμετέχοντες στη σημερινή ακρόαση και το επανειδήν. Ευχαριστώ. Sorry, I have to announce that the next meeting is coming when... Η επόμενη συνεδρίαση την Τετάρτη στις 23 Νοεμβρίου, ακρόαση για τα καινούργια και τα εφιστάμενα μέλη του Ελληνικού Συνεδρίου.